Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Θα σας διασκεδάσω λίγο που να έρθουν όλοι. Θέλω να σας καλωσορίσω λοιπόν 29 μέλη από τα κοινοβούλια των κρατών μελών, από 19 χώρες μαζί με υπαλλήλους των κοινοβουλίων συνολικά 72 συμμετέχοντες σε αυτήν την ανταλλαγή απόψεων για τον κύκλο του 2017 το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο είναι ένα κρίσιμο θα έλεγα σημείο πρέπει να συζητήσουμε τον κύκλο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Έχουμε τις συστάσεις τις οποίες υιοθέτησε τον Ιούλιο γιατί κάθε χώρα ξεχωριστά το Συμβούλιο και όπως γνωρίζετε τα κράτη-μέλη προετοιμάζουν τους προϋπολογισμούς τους και νομίζω ότι ελπίζω μέσα στις δημοσιονομικές ρυθμίσεις θα γίνουν σεβαστές αυτές οι συστάσεις αναχώρα. Έχει μεγάλη σημασία και για τα μεμονωμένα κράτη-μέλη, αλλά και αν θέλουμε να δούμε το θέμα με συνολικότερο τρόπο, σαν ευρωπαϊκό θέμα, γιατί βλέπουμε ότι ο ένας ή μία δημοσιονομική ρύθμιση σε μία χώρα επηρεάζει συνολικά τον προϋπολογισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και σε επίπεδο οικονομικό και σε επίπεδο αυστηρότερα δημοσιονομικό το θέμα αυτό με συνολικό ευρωπαϊκό τρόπο. Καλούμεθα τουλάχιστον να το κάνουμε. Όπως γνωρίζετε, Η έκθεση πρωτοβουλίας για τον κύκλο εξαμήνου 2017 βρίσκεται στην τελική φάση. Η συγητής μα είναι ο κ. ο οποίος μόλις μπήκε στην αίθουσα. Στόχος της παρούσας συζήτησης είναι να προχωρήσουν οι συζητήσεις πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία και να μπορέσουμε να ενημερώσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον κύκλο 2017 πριν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύσει την ετήσια έκθεσή της για την οικονομική ανάπτυξη και καθορίσει τις βασικές της προτεραιότητες για το 2018. Έχουμε πλέον δηλαδή ένα διτό στόχο. Από τη μία προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε και να αξιολογήσουμε τον κύκλο 2016-17 και να δούμε σε ποιο βαθμό έχουν <clears throat> ενσωματωθεί στις εθνικές λογικές ή κοινοτικές προτάσεις και από την άλλη προσπαθούμε να δώσουμε κάποιες συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για την ετήσια έκθεσή της για την ανάπτυξη και για τον επόμενο κύκλο του 18. Μια τεχνικής φύσεως παρατήρηση τώρα, να υπενθυμίσω στους συμμετέχοντες ότι είμαστε πολλοί στην αίθουσα και για να μπορέσουμε να διευκολύνουμε την συμμετοχή όλων των κοινοβουλίων των κρατών μελών, μόνο ένα μέλος ανασώμα θα μπορεί να πάρει το λόγο. Αν τυχόν τώρα μετά από τον πρώτο γύρο των παρατηρήσεων και των συζητήσεων υπάρξει χρόνος, τότε ίσως και κάποιο δεύτερο μέλος, εάν υπάρχει, μπορεί να ζητήσει το λόγο. Είδατε νομίζω την πρόταση εκθέσεως την οποία έχουμε προετοιμάσει. Υπάρχουν και οι τροπολογίες διαθέσιμες. Τώρα βρισκόμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα πλαίσια της φάσης αξιολόγησης των τροπολογιών και της προετοιμασίας των λεγόμενων συμβιβαστικών τροπολογιών οι οποίες ε, ομαδοποιούν και λαμβάνουν υπόψη τις διαφορετικές τροπολογίες ε, για να ενσωματωθούν στο τελικό κείμενο. Θα ήθελα να ξεκινήσω λοιπόν τη συζήτησή μας. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Χέκμαρκ. Θα μας παρουσιάσει την έκθεσή του ο κύριος Χέκμαρκ. Μετά θα δώσω το λόγο στους κοιόδης εισηγητές και φυσικά στους εκπροσώπους των κοινοβουλίων των κρατών μελών που το επιθυμούν. Θα προσπαθήσω να δώσω κατά προτεραιότητα το λόγο σε εκπροσώπους των κοινοβουλίων των κρατών μελών, εις βάρος αν θέλετε, των ε, μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο Γκούναρ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε, αγαπητοί συνάλλοι, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα απλά και μόνο να υπογραμμίσω ορισμένα ζητήματα τα οποία θεωρούμε και εγώ προσωπικά και οι υπόλοιποι συναδελφοί μου σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή οικονομία. Βέβαια δεν είναι και εύκολο, γιατί δεν υπάρχει και κάτι καινούριο ουσιαστικά εξορισμού. Είναι λίγο πολύ πράγματα τα οποία τα συζητάμε στα κράτη-μέλη, αλλά θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια σημαντικά σημεία παρόλα αυτά, για να καταλάβετε κι εσείς σε ποιο σημείο βρισκόμαστε έχουμε οικονομική ανάκαμψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι πολύ ευπρόσδεκτο φυσικά. Που θα μπορούσε να είχε έρθει και νωρίτερα, αλλά τέλος πάντων το σημαντικό είναι ότι έρχεται. Και αυτή η οικονομική ανάπτυξη, οικονομική ανάκαμψη, ε, αφήνει και κάποια περιθώρια για προσαρμογές. Δεν είναι όμως και πολύ δυνατή η ανάκαμψη αυτή, είναι αδύναμη, ακόμη τουλάχιστον. Είναι όμως ανάκαμψη που πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Είναι συνάρτηση και μιας ακραίας κομπής πολιτικής που τόνωνε τη ζήτηση της επενδύσης που θα ήταν πιο δύσκολο να έχει τα αποτελέσματα ε, τα ίδια μια πολιτική, πώς να την πω, φυσιολογική ας πούμε. Έχουμε και το στόχο των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Και στην έκθεσή μας λέμε ότι αν θέλουμε να υπάρξει σύγκληση των οικονομιών, των κρατών μελών, κάτι βέβαια πάρα πολύ σημαντικό, χρειάζεται σύγκληση και στο μέτωπο των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για να μπορέσουν να αναπτυχθούν οικονομίες. Αν δει κανεί ε, τι γίνεται σε επίπεδο κρατών μελών, ε, θα διαπιστώσει ότι οι επιδόσεις είναι διαφορετικές ανάλογα με το κράτος μέλος. Αν δει δε κανείς μόνο ομαδοποιημένα την κατάσταση, δεν μπορεί να αποκομίσει μια σωστή εικόνα. Παραδείγματος χάρη, αν όπως λέμε έχεις ε, στο ψυγείο το κεφάλι και τα πόδια στο φούρνο, η μέση θερμοκρασία είναι μια χαρά. Αλλά ούτε το κεφάλι ούτε τα πόδια είναι και σε καλή κατάσταση. Αυτό συμβαίνει αν συζητά κανείς ε, με βάση μοδοποιημένα μεγέθη στην ευρωπαϊκή οικονομία. Αντίθετα, θεωρώ πρέπει να εστιάζουμε στις διαφορές. Οι διαφορές αυτές υπογραμμίζουν άλλωστε και την ανάγκη για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, διότι είναι προφανές. Από όπου και αν προέρχεται κανείς, από όποια πλευρά του πολιτικού φάσματος, διαπιστώνει ότι κάποια κράτη-μέλη τα καταφέρουν καλύτερα από κάποια άλλα. Και αυτό βέβαια μπορεί να εξηγηθεί πάντοτε για, με κάποιους μη πολιτικούς λόγους. Γνωρίζω όμω ότι υπάρχει διαφορά. Α πούμε, στα κράτη-μέλη που δεν τα πηγαίνουν πολύ καλά, πολύ συχνά η εξήγηση που δίνεται είναι μη πολιτική. Προβάλλονται μη πολιτικοί λόγοι. Και το αντίθετο ισχύει στα κράτη-μέλη που τα πηγαίνουν καλά. Οι λόγοι που δίνονται δηλαδή είναι πολιτικοί κυρίω. Το θέμα είναι τι κάνουμε εκεί που δεν τα πηγαίνουμε τόσο καλά. Και σε αυτή την περίπτωση αυτό που επηρεάζει είναι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, είναι το πολιτικό θεματολόγιο. Και εκεί που τα πράγματα πηγαίνουν καλά, επίση η συγκυρία βοηθάει και οι συνθήκες βοηθούν, αλλά οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, η εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών βοηθάει ακόμη περισσότερο. Φαντάζομαι ότι αργότερα στο πλαίσιο τη συζήτηση θα ακούσετε ότι υπάρχουν διαφορετικέ απόψει από αυτού. Δηλαδή διαφορετικές απόψεις για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα των δημόσιων οικονομικών, των δραστικών μεταρρυθμίσεων. Εγώ όμως είμαι ξεκάθαρος στο πώς βλέπω τα πράγματα. Αν θέλουμε να ενεργούμε ως μια ισχυρή οικονομία σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον και να αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις της παγκόσμιας οικονομίας, τότε πρέπει οι επιδόσεις μας ομαδικά να είναι πολύ καλύτερες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άκει να δει κανείς τι γίνεται στον πλανήτη. Τα πράγματα έχουν αλλάξει. Άρδιν. Υπήρχαν πράγματα που κανείς δεν μπορούσε να τα φανταστεί πριν από 10 χρόνια. Και τώρα τα βλέπουμε μπροστά μας. Εγώ είμαι Σουηδός. Στη Σουηδία Έχουμε την εταιρεία των τηλεπικοινωνιών, την Ericsson, που για 10 χρόνια ήταν ένας αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη. Σήμερα όμως αμφισβητείται εντελώς η θέση της, για να μην πω ότι είναι στο 2 ή στο 3 στην κατάταξη πλέον, γιατί έχουμε την ε, Huawei, την κινέζικη εταιρεία, που είναι ένας πάρα πολύ ισχυρός ανταγωνιστής. Το ίδιο το βλέπει κανείς στην αυτοκινητοβιομηχανία, στην ε, διαστημική, ε, αεροδιαστημική, στην ιατρική. Παντού στον κόσμο βλέπουμε να αναδύεται ένα νέο ανταγωνισμό. Και αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη την ευρωπαϊκή οικονομία να είναι πιο ανταγωνιστική και ισχυρότερη, να μπορεί να αναπτυχθεί καλύτερα, περισσότερο. Και αυτό πρέπει να το πετύχουμε από κοινού, όλοι μαζί. Όμω, για να αυξηθεί ο μέσο όρο, θα πρέπει εκεί που είμαστε κάτω από το μεσόρο να τα πάμε καλύτερα. Δεν είναι και τόσο εύκολο αυτό, είδε από πολιτική πλευρά. Ε, υπάρχουν πολλέ πολιτικέ προκλήσει. Αλλά και από οικονομικής μαθηματικής πλευράς δεν είναι και τόσο εύκολο. Δηλαδή κάποιες φορές είναι πιο δύσκολο να ξεπεράσει κανείς το μεσόωρο ή να προσπαθήσει να τον φτάσει από ότι να τα καταφέρει καλύτερα όντας ήδη πάνω από το μεσόωρο. Πάντως πρέπει να έχουμε ένα κοινό στόχο. Μια δυνητική ανάπτυξη, τουλάχιστον δυνητική λέω, της τάξης του 3% όλες οι οικονομίες μας θα πρέπει να είναι σε θέση να έχουν αυτή την επίδοση της ανάπτυξης του 3% των τριών ποσοστιών μονάδων. Αν το πετύχουμε, αν έχουμε αυτή την ε, σύγκληση προς τα πάνω, να μην είναι λέει, κανείς κάτω από το μέσο όρο αν θέλετε, που βέβαια μαθηματικώς αυτό είναι ανέφικτο γιατί πρέπει να υπάρχει ένας μέσος όρος, πάντα πρέπει και θα υπάρχει ένας μέσος όρος, αλλά αν καταφέρουμε να αυξήσουμε το επίπεδο της οικονομίας πάνω από το μέσο όρο, τότε θα είναι πολύ πιο υψηλός ο μέσος όρος αυτός. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για όλα τα κράτη-μέλη και για την ευρωπαϊκή οικονομία. πρόκληση όμως είναι οι σημερινέ οικονομίε να έχουν ακόμη καλύτερε επιδόσεις. Χωρίς να επαναπαύονται. Μπορεί να νομίζουν ότι τα πηγαίνουν καλά και είναι στο απειρόβλητο, αλλά δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Στη χώρα μου είχαμε τις τελευταίες, τα τελευταία 10-15 χρόνια καλές επιδόσεις, αλλά και εμείς δεχόμαστε επιθέσεις και εμείς αντιμετωπίζουμε προβλήματα και πρέπει να ανθέξουμε στις δυσκολίες. Ελπίζω αυτή η έκθεση που ελπίζω να γίνει και κοινή απόφαση να εστιάσει σωστά. Εμείς θέλουμε ε, να εστιάσουμε στη δημοσιογραφική σταθερότητα, αλλά οι απόψει μα διαφέρουν. Επίση, ό,τι αφορά τι διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εσωτερική αγορά δηλαδή και άλλα. Και εκεί πρέπει να συμφωνήσουμε. Και επίση θα πρέπει να εφαρμοστούν οι μεταρρυθμίσει και στι εθνικέ οικονομίε. Η σύγκληση οικονομική και κοινωνική σημαίνει ότι χρειάζεται σύγκληση και στις διδροτικές μεταρρυθμίσεις και στη δημοσιονομική σταθερότητα. Πρέπει να έχουμε αυτό το κοινό στόχο. Τουλάχιστον 9% αύξηση της ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονομίας. Για να μπορέσουμε να αναπτυχθούμε καλύτερα και να βρεθούμε σε καλύτερη θέση απέναντι στους ανταγωνιστές και να πάρουμε στα χέρια μας τα ενία κάτι που είναι πολύ σημαντικό και φέρνει ευημερία και πλούτο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Uh, Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή μας. Είναι εκπρόσωπος του ΕΛΚΑ, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Θα δώσω τώρα το λόγο στον σκιώδη εισηγητή που είναι εκπρόσωπος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, τον κύριο Σίλβα Περέιρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχάς, θέλω να καλωσορίσω όλους τους συναδέλφους που ήρθαν εδώ από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Σας καλωσορίζω θερμά στην Επιτροπή μας. Δράτομαι επίσης της για να ευχαριστήσω και τον εισηγητή μας, τον κύριο Χέκμαρκ. Είχαμε πολύ επικοδομητικές συζητήσεις ε, για τις οικονομικές πολιτικές ε, στο πλαίσιο της Ευρωζώνης. Το πρώτο σημείο στο οποίο θα ήθελα να επιμείνω είναι πως η ευρωπαϊκή οικονομία και δι η οικονομία της Ευρωζώνης επιτέλους παρουσιάζει σημάδια ανάκαμψης. Κάτι το οποίο πρέπει να μας χαροποιεί. Ταυτόχρονα βέβαια παραμένει το γεγονός ότι είναι αδύναμη η ανάκαμψη αυτή που παρατηρούμε. Υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα και πολύ είναι κίνδυνη και ιδίως πολιτικού χαρακτήρα. Επίσης η οικονομική αυτή ανάκαμψη δεν είναι καθόλου ισομερής αν θέλετε, είναι άνηση. Είναι μια ανισότητα που οφείλεται στις μεγαλύτερες, στις αυξανόμενες ανισότητες και αποκλίσεις που βλέπουμε στα χρόνια τα τελευταία να διωγγούνται. Και γι' αυτό το λόγο, αντί να θριαμβολογούμε για το πόσο καλύτερα πηγαίνουν τα πράγματα, αυτό που θα έπρεπε να κάνουμε στην παρούσα φάση είναι να επιμένουμε στο ότι εξακολουθεί να απαιτείται μια πολιτική αντίδραση σε ό,τι αφορά την οικονομική και δημοσιονομική πολιτική, ούτω ώστε να αντιμετωπίσουμε κατά μέτωπο τις προκλήσεις και να δρομολογήσουμε και πάλι το ευρωπαϊκό όραμα. Να ξαναπροσδεθούμε στο άρμα της σύγκλησης. Αυτές οι διωγγούμενες ανισότητες και αποκλείσεις μεταξύ των κρατών μελών που χειροτέρεψαν τα τελευταία χρόνια δεν είναι μόνο οικονομικό πρόβλημα αλλά και πολιτικό πρόβλημα για το μέλλον του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Υπάρχουν επενδυτικά κενά και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. στο σχέδιο Juncker συμφωνήσαμε να επιμηκυνθεί. Και αυτό είναι θετικό. Δεν θα λύσει όμως όλα τα προβλήματα. Θα είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει μια δίκαιη γεωγραφική κατανομή, κάτι το οποίο είναι απαραίτητο αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τις ασυμμετρίες και τις, ασυμμετρίες και τις ανισότητες που υπάρχουν. Αυτό το οποίο χρειάζεται, τι είναι λοιπόν. Φυσικά και χρειάζεται νομισματική πολιτική που να στηρίζει την ανάπτυξη και στο μέλλον όπως και τώρα και ιδίως μιλώντας για την Ευρωζώνη. Θα χρειαστούμε όμως ακόμη συμπληρωματικά και δημοσιονομική πολιτική μέτρα δημοσιονομικά που θα στηρίζουν και αυτά την ανάπτυξη. Δημοσιονομική πολιτική η οποία αξιοποιεί την ευελιξία που προβλέπουν οι κανόνες μας για να στηρίξει την οικονομία, όχι να την στραγγαλίσει. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το 2017, πρόσφατα μάλιστα, εξέδωσε μια ανακοίνωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά τη και είπε ότι είναι μετεριοπαθώς επεκτατική και οι χώρες με μεγαλύτερα δημοσιονομικά περιθώρια θα έπρεπε να κάνουν μια παραπάνω προσπάθεια για να βελτιωθεί συνολικά η ζήτηση και να υποστηριχθεί η ανάπτυξη. Αυτό που βλέπουμε όμως είναι πλήρης απουσία ε, αυτού του πράγματος. Βλέπουμε αντίθετα ουδέτερη, στην καλύτερη περίπτωση, δημοσιονομική πολιτική. Άρα, μπορούμε να μιλήσουμε διαμακρών για ανάπτυξη και σύγκληση, και να προωθήσουμε όσες ε, διαφορετικές βερσιών του σχεδίου Juncker θέλετε. Μπορούμε να προωθήσουμε τις διαφορετικές μεταρρυθμίσεις για να λύσουμε τα προβλήματα. Συζητώντας όμως για πολύ καιρό τι θα πει διαρθρωτική πολιτική. Τι πρέπει να κάνουμε όμως εμείς τελικά στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Πρέπει να συζητήσουμε για τη δημοσιονομική πολιτική και να συζητήσουμε κατά πόσον αυτή η δημοσιονομική πολιτική που έχουμε είναι αρκετά ισχυρή ώστε να στηρίξει το δυναμισμό της οικονομίας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Αυτή είναι η μείζων ανησυχία των σοσιαλιστών και δημοκρατών στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης. Και ελπίζω ότι στο πέρας αυτής της ε, συζήτησης, της έκθεσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ενώσει τη φωνή του στις φωνές των άλλων θεσμικών οργάνων που ζητούν μια δημοσιονομική πολιτική που θα είναι μετριοπαθώς επεκτατική. Το λιγότερο δεν είναι και κάτι υπερβολικό πιστεύω ως αίτημα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Οντόνελ. Από την Βουλή της Ιρλανδίας. Παρακαλώ. Thank you, Chairman. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε καλοδεχούμενη έκθεση και όσον αφορά τις συστάσεις για την Ιρλανδία, πολλές από αυτές έχουν ήδη υλοποιηθεί. Σήμερα κατατίθεται ο προπολογισμό, οπότε αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο Υπουργό ε, των Οικονομικών ανακοίνωσε τον προπολογισμό. Κάποια πράγματα στις συστάσεις αναχώρα, το 1,5 δισεκατομμύριο το Ταμείο Ανάγκης, ε, θα περικοδοτηθεί με ένα μισθής και άλλο ένα δις κάθε χρόνο. Όσον αφορά την ε, ανεργία, τα τελευταία 19 τρίμηνα είχαμε ε, μείωση της ανεργίας. Ε, έχουμε 6% ανεργία αυτή τη στιγμή, σχεδόν πλήρη απασχόληση. Είχαμε 15% ανεργία το 2008-2009, οπότε έχουμε κάνει μεγάλα βήματα στην πλευρά των επενδύσεων. Οπωσδήποτε όταν ξεκίνησε η οικονομική κρίση δεν είχαμε καμία επιλογή παρά να μειώσουμε τις δαπάνες. Μέχρι το 2021, σε σύγκριση με το 2015, αναμένουμε να διπλασιάσουμε τις ε, επενδύσεις από 3,7 δις το 2015 θα πάει σχεδόν 8 δισεκατομμύρια το 2021. Το 2018 θα έχουμε μία αύξηση 800 εκατομμυρίων, 17% αύξηση δηλαδή, κάτι το οποίο νομίζω είναι πολύ θετικό και πραγματικά θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει, δηλαδή να ρίξουμε λεφτά σε επενδύσεις, συγκεκριμένα στον τομέα της στέγασης ε, που αναφέρεται στην έκθεσή σας δύο στοιχεία όσον αφορά τις ε, κοινωνικές ε, κατοικίες αλλά και τον ιδιωτικό τομέα. Ε, το τρέχον έτος έχουμε 1,83 δισεκατομμύρια για την κοινωνική στέγαση για να δημιουργηθούν σχεδόν 4.000 νέες κατοικίες. Δημιουργούμε ένα συγκεκριμένο ταμείο που θα δίνει πρόσβαση στην χρηματοδότηση για να χτιστούν ιδιωτικές ε, κατοικίες. 750 ε, εκατομμύρια ρίχνουμε εκεί. Και βεβαίως ε, έχουμε, όπως σας είπα, το θέμα της προσφοράς και όσον αφορά το όλο θέμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων στις ε, τράπεζες είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ειδικά για τα άτομα τα οποία θέλουν να παραμείνουν στα σπίτια τους ε, έχουμε ένα ειδικό ε, μέσο για τα στεγαστικά δάνεια και εν ολίγης αναμένουμε ε, ότι θα επιτύχουμε το μεσοπρόθεσμο στόχο του 0,5% διαρθρωτικό έλλειμμα το 2018 επιβεβαιώθηκε στο σημερινό προϋπολογισμό από τον Υπουργό Οικονομικών και αναμένουμε ίσως και λυσμένο προϋπολογισμό προσεχώς και θα περάσουμε σε πλεόνασμα. Τα επίπεδα του χρέους γενικώ ε, μειώνονται και φαντάζεστε ότι ε, έχουμε μεγάλο ρυθμό ανάπτυξης. Ε, το 2007 αναμένουμε 4,3, το 2018 3,5% είναι νομίζω βιώσιμη ρυθμή ανάπτυξης ε, και αντιμετωπίζονται έτσι οι περισσότερες συστάσεις που έγιναν προς την Ιρλανδία. Για εμάς το Brexit είναι τεράστιο ζήτημα και Θα ήθελα εγώ να ευχηθώ καλή επιτυχία στις ε, συζητήσεις. Γιατί είμαστε μικρή εξαγωγική οικονομία και έχει μεγάλη σημασία για μας αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο εκπρόσωπος από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Κύπρου. Ε, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως γνωρίζετε, η Κύπρος ολοκλήρωσε με επιτυχία το, το πρόγραμμα προσαρμογής εντός του 2016. Έγιναν αρκετές μεταρρυθμίσεις στα πλαίσια εκείνου του προγράμματος, όπως η καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού στη δημόσια υπηρεσία, μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος και πολλά άλλα. Ήδη βλέπουμε αυτά τα θετικά αποτελέσματα. Ε, σήμερα που μιλάμε έχουμε μάλλον εδώ και δύο-τρία χρόνια ίσως κελισμένο προϋπολογισμό πάμε και για ένα σχετικά μεγάλο πλεόνασμα εντός του 2017 πέραν του 1% του ΑΕΠ, όχι πρωτογενές πλεόνασμα, δημοσιονομικό πλεόνασμα. Το πρωτογενές πλεόνασμα είναι ακόμα μεγαλύτερο και απολαμβάνουμε και ψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Εντός του 2016 ήταν γύρω στο 2,8% φέτος προβλέπεται να ξεπεράσουμε ή να είμαστε κάπου στο 3,5% αυτή την πορεία να μένουμε και για, τα, και για το 2018. προϋπολογισμός και πάλι αφορά ένα ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, μάλλον ένα προϋπολογισμό που εκτιμώ ότι και πάλι θα έχουμε πλεόνασμα με συντηρητικές προβλέψεις πάντοτε. Α, όσον αφορά τις ειδικέ συστάσεις, συμφωνούμε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ήδη έχουν προχωρήσει κάποια πράγματα από τότε. Για παράδειγμα, έχουμε ήδη ψηφίσει το, την εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας που θα είναι μια καθολική κάλυψη για όλον τον πληθυσμό και είναι μία από τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Α, κάποιες άλλες μεταρρυθμίσεις πρέπει να κατανοήσουμε ότι ενδεχομένως δεν έχουν την κοινωνική και πολιτική πλειοψηφία όπως για παράδειγμα η, η ιδιωτικοποίηση οργανισμών κοινή ωφελία, έστω αν κάποιοι συμφωνούμε, μπορεί να μην αποκτήσουν αυτή την πλειοψηφία. Προσπαθούμε να βρούμε όμως ε, συγκεκριμένες ε, συνενέσεις. θέλω να πω πως και οι προβλέψεις των οίκων αξιολόγησης για τα επόμενα τρία χρόνια λένε ακριβώς ότι η Κύπρος μπορεί να πετύχει πλεονάσματα και υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης ταυτόχρονα, άρα ίσως ένα δίλημα που μα απασχολεί συχνά κατά πόσο είμαστε υπέρ της ανάπτυξης ή της λιτότητας, να, να μην είναι ένα αυτό καθ' αυτό πραγματικό ε, δίλημα. Μπορούμε να καταφέρουμε μέσα από ανάλογες μεταρρυθμίσεις ε, τον στόχο για ισοσκελισμένους προπολογισμού, ικανοποιητική ανάπτυξη, μείωση της ανεργίας, Έχουμε όλα αυτά, μπορούμε να τα δούμε. Πλην όμως πρέπει, πιστεύω, να γίνει κατανοητό πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να είναι απλά ένας οργανισμός που επιβάλλει μεταρρυθμίσεις στα κράτη-μέλη. Πρέπει να μεταρρυθμιστεί και η ίδια. Γιατί η ίδια ιδιότητα του κράτους μέλους μπορεί να έχει πλεονεκτήματα, ιδίω στην Ευρωζώνη υπάρχουν όμως και σημαντικά μειονεκτήματα. Το ότι δεν υπάρχει η αυτόνομη νομισματική πολιτική. Γνωρίζουμε ότι η Ευρωζώνη δεν είναι μια τέλεια νομισματική ένωση, είναι μια ατελής νομισματική ένωση για την οποία πρέπει να εργαστούμε προς και εκείνη την κατεύθυνση. Α, σήμερα η οίκοι αξιολόγηση και οι αγορές γνωρίζουν ότι σε περίπτωση κρίσης δεν θα μπορεί το κάθε κράτος μέλος να ασκήσει την δική του αυτόνομη νομισματική πολιτική. Αυτό φαίνεται και στα επιτόκια δανεισμού στις αγορές. Όταν δημιουργήθηκε η Ευρωζώνη είχαμε μια σύγκληση επιτοκίων. Τώρα έχουμε μια τεράστια απόκληση επιτοκίων. Άρα εκείνο το οποίο θα ήθελα να πω και σαν Ευρωπαίος πολίτης το λέω αυτό που θέλω να πετύχει το, το ευρωπαϊκό όνειρο να είμαστε μια δυνατή ένωση με επιρροή στον πλανήτη είναι ακριβώς ότι πρέπει να δούμε και τα θεμέλια της ίδιας της νομισματικής ένωσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Uh, uh, Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Βάλη, σκιώδης εισηγητής από την ομάδα EFTD έχει το λόγο. Ε, εγώ εδώ και τρία χρόνια ασχολούμαι με το θέμα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και πολύ συχνά έχουμε εντελώς διαφορετικές απόψεις για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να προχωρήσουμε. Η τελευταία παρέμβαση που έγινε πριν από μένα από τον Κύπριο συνάδελφο το υποδεικνύει αυτό. Υπάρχουν λοιπόν μεταρρυθμίσεις σημαντικές οι οποίες πρέπει να γίνουν στο εσωτερικό της Ευρωζώνης και αυτό πρέπει να είναι μια προτεραιότητα για μας. Η ανάπτυξη η οποία έχει υπάρξει μέχρι τώρα θα έλεγα οφείλεται ε, στις τεράστιες προσπάθειες που έχουμε κάνει σε οικονομικό επίπεδο και το 10% μόνο σε πολλές μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει σε δημοσιονομικό επίπεδο. Πολλές φορές ε, έχουν ε, υπάρξει σαν παράδειγμα καθόλου δημοφιλείς πολιτικές απαξίωσης ουσιαστικά των μισθών, των συντάξεων κτλ. Συνεπώς λοιπόν θα πρέπει να είμαστε ειλικρινεί και να δούμε τι ακριβώς ανάγκες έχουμε, να δούμε τι ανισότητες και ελλείψεις ισορροπίας υπάρχουν στο εσωτερικό της ζώνης ευρώ. Η διαδικασία Micro Balance Procedure, ή σαν παράδειγμα, είναι ένα σημαντικό πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να προσπαθήσουμε να το επιλύσουμε Χώρες όπως η Ολλανδία και η, η Γερμανία παραβιάζουν τέτοιου είδους κανόνες και δημιουργούν ε, μια έλλειψη ισορροπίας η οποία επηρεάζει συνολικά την Ευρωζώνη. Μια πρόταση λοιπόν όπως αυτή των ε, μεταφορών από τις περιφερειακές ε, περιοχές στο κέντρο είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει στην δημιουργία ενός ε, Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σταθερότητας, το οποίο όμως δεν θα ήταν και πάρα πολύ δημοκρατικό με τον τρόπο που θα μπορούσε να λειτουργήσει για να σταθεροποιήσει το εσωτερικό της ζώνης ευρώ. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να δούμε ποιες είναι οι προτάσεις οι οποίες έχουν αρχίσει να μορφοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε επίπεδο Eurogroup πιο συγκεκριμένα και να προσπαθήσουμε να κατευθύνουμε κατά κάποιο τρόπο το ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το οποίο να μην είναι τόσο άμορφο όσο είναι τώρα και να μην είναι τόσο γερμανικό όσο είναι τώρα. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αφήσουμε τη λιτότητα ως αυτοσκοπό και να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε μια Ευρώπη η οποία να λειτουργήσει με ειλικρίνεια, για την επίτευξη των οικονομικών στόχων. Στην έκθεση αυτή κάτι τέτοιο δεν φαίνεται, δεν το είδα ούτε στο παρελθόν. Το θέμα αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα έλεγα μας έχει απασχολήσει στο Ευρωπαϊκό Γενοβούλιο. Οι προτάσεις τις οποίες θα κάνουμε όμως θα πρέπει να είναι εφαρμόσιμες και δημοκρατικές και όχι το αντίθετο γιατί αλλιώς δημιουργούνται ανησυχίες όπως αυτές που ακούσαμε από τους προηγούμενους συναδέλφους. Ε, έχουμε αρνητικές συνέπειες στις δημοσιονομικές πολιτικές που ακολουθούμε, όπως ε, η απαξίωση των μισθών. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε μεταρρυθμίσεις, αλλά με ειλικρίνεια να δούμε ποιες είναι οι αδυναμίες της Ευρωζώνης, να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σωστά τη δημόσια δαπάνη, γιατί η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα τα προβλήματα που έχουμε παραμένουν όπως και στο παρελθόν. Είναι προβλήματα διαρθρωτικού τύπου. Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε στην κρίση να ξαναγυρίσει να μας χτυπήσει με τα ίδια παλαιά μέσα. Ευχαριστώ πολύ. Από την Ιταλική Γερουσία τώρα, εκπρόσωπος της Ιταλικής Γερουσίας. Thank you very Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ με τον εισηγητή ότι η οικονομική ανάκαμψη είναι κάτι το καινούριο για την Ευρωζώνη και συμφωνώ ότι η οικονομική ανάκαμψη εξακολουθεί να είναι ασθενής και εύθραυστη. Ειδικά ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης, εάν το συγκρίνουμε με το παρελθόν δεν είναι πολύ ικανοποιητικό. Βεβαίως μπορούμε να πούμε ότι έχουμε οικονομική ανάκαμψη αλλά δεν έχουμε κάποια πορεία ανάπτυξης, έναν μηχανισμό δηλαδή που θα μπορεί να συντηρείται μέσω μιας τέτοιας ε, οικονομικά επεκτατικής πολιτικής. Βεβαίω τα αδύναμα σημεία είναι οι επενδύσεις που είναι ακόμα πολύ χαμηλές στην Ευρωζώνη και η παραγωγικότητα που είναι πολύ χαμηλή. Αυτές είναι οι μεσομακροπρόθεσμες ε, τάσεις ε, που δικαιολογούν ε, το γιατί δεν είμαστε πολύ ικανοποιημένοι. Και προσέθεσε ο εισηγητής πως έχουμε αποκλίνουσες αποδόσεις των διαφόρων χωρών, κάτι το οποίο είναι μια μεγάλη ενισχύ. Οπότε, μία πρόταση είναι το πώς θα βελτιωθούν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στο εθνικό επίπεδο. Στην περίπτωση της Ιταλίας υπάρχουν στις συστάσεις ε, για την χώρα για το 2016 και για το 2017 κάποια πράγματα που πρέπει να γίνουν. Κάναμε πολλά πράγματα, επιτύχαμε ουσιαστική πρόοδο σε πολλά μέτωπα, αλλά ακόμα κάποια άλλα πρέπει να γίνουν. Αλλά αυτό το οποίο πρέπει να τονίσουμε πολύ περισσότερο είναι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στο επίπεδο της Ευρωζώνης. Αν δείτε τις συστάσεις για την Ευρωζώνη το 2016, βλέπουμε τις ίδιες συστάσεις και το 17. Και όπως λέτε, δεν υπάρχει τίποτα το καινούριο. Ε, τίποτα καινούριο σε δύο μέτωπα. Πρώτα απ' όλα η δημοσιονομική στάση. Αυτό δεν είναι πολύ γιατί θέλετε, ε, θέλω πιο επεκτατική τέτοια στάση ή λιγότερη. Γιατί χρειάζεται μια προσέγγιση η οποία δεν θα είναι μόνο στοχευμένη σε εθνικό επίπεδο, αλλά με κάποιον τρόπο θα πρέπει να ορίζει το τι απαιτείται σε επίπεδο ευρωζώνης. Και βεβαίως αυτή ακριβώς ε, η στάση είναι κάτι το οποίο είναι αφηρημένο. Η Κομισιόν έκανε μια πρόταση πέρσι, έκανε κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις οι οποίες απορρίφθηκαν. Οπότε εγώ θα τόνιζα ότι πρέπει να το καθορίσουμε πολύ καλύτερα γιατί είναι κάποια μέσα συμπληρωματικά για να διατηρηθεί αυτός ο ρυθμός ανάπτυξης. Και δεύτερον, οι τάσεις των επενδύσεων στην Ευρωζώνη ε, είχαν πολύ θετικές εμπειρίες το σχέδιο Juncker, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι πολύ καλό ως μια δοκιμή μικρής κλίμακας. Θα πρέπει λοιπόν η ίδια λογική να εφαρμοστεί σε μεγαλύτερη κλίμακα. Η πρότασή μου είναι λοιπόν να περιλάβουμε σε αυτήν την έκθεση πολύ περισσότερο τις προτάσεις αυτές. Πώς θα βελτιωθούν δηλαδή οι συστάσεις και ο ρυθμός εφαρμογής τους για να μην ξαναδιαβάσουμε το 2018 τις ίδιες συστάσεις που διαβάζουμε τα τελευταια δυο δύο-τρία χρόνια. Αυτό έχω εγώ να προτείνω και σύμφωνο ότι η ανάκαμψη είναι θετική αλλά πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα για να αυξηθεί ο ρυθμός ανάπτυξης ε, της, ε, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Σας ευχαριστώ ο κύριος Μπαλαούρας ε, από τη Βουλή των Ελλήνων. Έχετε το λόγο. μικρόφωνο σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Άκουσα με πάρα πολύ προσοχή και τους ε, δύο πρώτους συγητές. Ε, ο πρώτος μίλησε για μία ανάκαψη η οποία είναι ασθενής, αλλά υπάρχει. Εγώ θα έλεγα ότι θα έπρεπε να σημειωθεί ότι άρχισε πάρα πολύ ακόμα και αυτή η ασθενής ανάπτυξη να έρθει. Πάρτε για παράδειγμα τις Ηνωμένε Πολιτείε. Μαζί μπήκαμε στην κρίση, έχουν βγει τώρα περίπου τέσσερα χρόνια, η Ευρώπη ακόμα παραδέρνει σε μια ε, ανάκαψη με πολύ ερωτηματικά με πολλά ερωτηματικά. Ε, ο δεύτερος ηγητής από το Σοσιαλιστικό Κόμμα, ο κύριος Περέιρα, ε, μίλησε ότι αυτή, αυτή η πορεία της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης θα προκαλέσει πολιτική αντίδραση. Και θέλω να πω ότι πράγματι, επειδή τα προβλήματα είναι πολιτικά και δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, θα υπάρξουν αντιδράσεις και ήδη τις βλέπουμε τις αντιδράσεις. Σε μια ε, σειρά από κράτη βλέπουμε αντιδράσεις οι οποίες οδηγούν έξω από μια δημοκρατική νομιμοποίηση κάποιες πολιτικές θέσεις και εκφράσεις. Πάμε στο, στα διατάφτα, τα οποία θέλω να τα συνδέσω τα οικονομικά πράγματα με τα πολιτικά το σύμφωνο σταθερότητας. Αν υποθέσουμε ότι παρήγαγε κάτι, σήμερα φαίνεται ότι δεν μπορεί να παράξει τίποτα. Τέλειωσε. Είναι σαν μια θηλιά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό το συνδέω με την ακροδεξιά, με το αυγό του φιδιού που έχει βγει πια και αγκαλιάζει πολλά κράτη και λαούς. Πρέπει να αντικατασταθεί από ένα σύμφωνο ανάπτυξης και εργασίας. Για παράδειγμα, να σας πω ότι στο καταστατικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δεν υπάρχει πουθενά η λέξη εργασία, απασχόληση. Μιλάει για πληθωρισμό, μιλάει και για ισορροπία στην νοσματική σφαίρα. Τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Σήμερα λοιπόν το αποτέλεσμα είναι να έχουμε ανισότητες περιφερειακές και κοινωνικές έντονα μεγάλες, ακόμα και εντό των κρατών, ανεργία, ιδιαίτερα στους νέους και δεν εννοούμε την Ελλάδα που η ανεργία ήταν πάνω από 60% ας πάρουμε άλλα κράτη, ας πάρουμε την Ισπανία, ας πάρουμε ε, τα κράτη του Νότου, ας πάρουμε και ορισμένα κράτη του Βορρά. Η ανεργία των νέων είναι σε δυσθεώρητα επίπεδα. Δεν μας προβληματίζει άρα γι' αυτό. Και τέλος έχουμε αυτή που είπαμε προηγουμένως περιορισμένη ανάπτυξη γιατί αντιμετωπίζεται η Ευρώπη αλλά κάρτ. Κάποιες δυνάμεις, ιδιαίτερα οι μεγάλες δυνάμεις ευρωπαϊκές, την αντιμετωπίζουν αλλά κάρτ. Άκουσα και όχι μόνο σήμερα και σήμερα ότι να προχωρήσουμε σε μεταρρυθμίσεις μεταρρυθμίσεις. Μια λέξη η οποία πρέπει να, την, να της δώσουμε ε, περιεχόμενο. Μετα, μεταρρυθμίσεις προς τι. Μεταρρυθμίσεις γιατί και για ποιους. Αν δεν τα προσδιορίσουμε αυτά τα πράγματα θα είναι μια λέξη η οποία είναι παραπλανητική. Και έχει γίνει πάρα πολλές φορές ε, παραπλανητική για όλους τους λαούς. Και όχι μόνο για τους λαούς που υποφέρουν σαν τον ελληνικό λαό. Επομένως, η θέση η δικιά μου, η θέση η δικιά μας που εκφράζουμε, μια, εκφράζουμε πολιτικές δυνάμεις που έχουν άλλο, ένα άλλο όραμα ευρωπαϊκό για μια, καλύτερη πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους λαούς να είναι πολύ καλύτερα να ξεφύγουν αυτή τη μέγενη της λιτότητας και της ανεργίας και να πάνε σε άλλα πράγματα. Προτείνουμε λοιπόν να υπάρξουν κρατικές επενδύσεις. Έχει ξεχαστεί αυτό το, το πράγμα. Επενδύσεις σε χώρες ιδιαίτερα που έχουν ανάγκη. Να υπάρξει εκδημοκρατισμός και διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί να υπάρχει το Eurogroup και να αποφασίζει για τη ζωή κυριολεκτικά των ανθρώπων χωρίς να έχει νομιμοποίηση. Δεν υπάρχει όργανο που λέγεται ε, ε, Eurogroup. Και όμως αποφασίζει για για χιλιάδες και εκατομμύρια ανθρώπους. Επομένως, επίσης θα πρέπει να κοιτάξουμε τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένας προϋπολογισμός που προσφέρει στη σύγκληση που είναι μια θέση, μια αρχή από το καταστατικό της ε, η δημιουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, αγαπητοί συνάδελφοι, η Λευκή Βίβλος και η έκθεση των πέντε προέδρων δεν έχουν συγκεκριμένε προτάσει. Θα μπορούσαμε να το πούμε σαν μια έκθεση ιδεών. Ενδιαφέρουσα. Αλλά συγκεκριμένε προτάσει για εκδημοκρατισμό και ανάπτυξη. Με τη συμμετοχή όλων. Βιώσιμη λοιπόν δίκαιη ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον. Ενδυνάμωση της νομοθεσίας, κύριε Πρόεδρε, για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος και της φοροδιαφυγής και του λαθρομπορίου. Αυτά πρέπει να, τα πάρει μπροστά της Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι το μόνο το ε, κάθε κράτος ξεχωριστά. Τέλος, προστασία των εργαζομένων με μήνυμους μισθούς, με συλλογικές συμβάσεις. Από πουθενά δεν προκύπτει ότι όπου υπάρχουν εργασιακές σχέσεις ελαστικές οδηγούν στην ανάπτυξη. Επομένως λέμε όχι στη λιτότητα, όχι σε ανάπτυξη για όλους. Ευχαριστούμε. Θα βάλω το χρονόμετρο από εδώ και πέρα. Τρία λεπτά ο καθένας. Η Γκαμπριέλα Κρέτσου από τη Ρουμανία, τη Γερουσία. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητοί συνάδελφοι. Θέλω να τονίσω κάποια πολύ ευαίσθητα ε, λεπτά πολιτικά ζητήματα. Η έκθεση προτείνει ή μάλλον λέει ότι είναι κάτι διαφορετικό το κράτος μέλος της Ευρωζώνης ε, και το κράτος μέλος που δεν ανήκει στην Ευρωζώνη με οικονομικές και μοσμετικές πολιτικές διαφορετικές ε, και με κάποιο είδους φανταστικά σύνορα. Πιστεύουμε ότι είναι μια πολύ ασφαλμένη προσέγγιση δεν θα μπορέσουμε αυτόν τον τρόπο ούτε να καταλάβουμε ούτε να λύσουμε το πραγματικό πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποια επιχειρήματα. Έχουμε μια νέα αγορά. Με τις τέσσερις ελευθερίες, για τις οποίες είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι. Μόνο η Δανία έχει μια εξαίρεση, ένα opt-out για το ευρώ. Η χρήση του ευρώ στις εγχώριες συναλλαγές είναι της τάξης 5-70%. Πολύ ψηλά ποσοστά σχεδόν σε όλες τις χώρες. Εμπόριο. Κατά 70% γίνεται στην ενή αγορά. Οι διεθνείς ε, εταιρείες, ευρωπαϊκές εταιρείες, πολυεθνικές δεν έχουν σύνορα. Χρησιμοποιούν μάλλον έχουν δραστηριότητε σε κράτη-μέλη που δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη. Και έχουμε προσπαθήσει να έχουμε έναν οικονομικό και νομισματικό συντονισμό μεταξύ μας. Η δημοσιονομική αυτονομία έχει κάποια όρια. Οι εθνικέ τράπεζε. δεν έχουν αρκετά εργαλεία στη διάθεσή τους για να μπορέσουν να τερματίσουν έναν ισχυρό ρόλο στι εθνικέ νομισματικέ πολιτικέ. Οι κυβερνήσει έχουν περιορισμού. Και το έχουμε καταλάβει αυτό. Οικειό, δημοσιονομικά ελλείμματα περιορισμένα το ευρωπαϊκό εξάμεινο κτλ. κτλ. Στάση αναχώρα. Όταν μιλάμε λοιπόν για ευρωζώνη και μη ευρωζώνη, αν χρησιμοποιούμε αυτούς τους όρους, υπονομεύουμε την αλληλεγγύη, υπονομεύουμε την ενότητα. Και τελικά τροφοδοτούμε τους ευρωσκεπτικιστές και τους λαϊκιστές που κάνουν τη διάξη μεταξύ αυτών, λένε αυτοί και εμείς. Και ταυτόχρονα που κρύπτουμε τα δύο βασικά προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θεσμικό που είναι ακριβώς το ευρώ, δηλαδή το κοινωνόμισμα να γίνει πραγματικά κοινό, ενιαίο. Και υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα ουσιοδέστατο που είναι η ανισότητα. Η πρότασή μας δεν είναι. Μάλλον είναι να μην ξεχνάμε να ζητούμε από την Κομισιόν να κάνει μία αναθεώρηση του Μεσονικού Συμφώνου. Πέντε χρόνια πάνε από τότε που τέθηκε σε ισχύ. Χρειάζεται αυτή η αξιολόγηση. Δεύτερον, για μας, όλους μας. Υποχρεωτικά θα πρέπει να το σκεφτούμε το θέμα. του σχέδιου Γιούγκερ. Τι ξεκίνησε με αυτό το σχέδιο Γιούγκερ. Οι άμεσε επενδύσει. οι ξένε άμεσες επενδύσεις ουσιαστικά αντικαταστάθηκαν από κίνητρα και έγκυα τα οποία, ε, επενδύσει τέλο πάντων, ε, οι οποίες ουσιαστικά καλύπτονται με δημόσια χέγγια αλλά γίνονται από το ιδιωτικό τομέα. Thank you very much. Um, ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τοσκάνη από την Περιφερειακή Βουλή της Γερμανίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και για την δυνατότητα που μας δίνεται να μπορούν να εκφραστούν εδώ τα εθνικά κοινοβούλια. Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάστηκε αυτή την έκθεση. Θεωρώ ότι βλέπει τα πράγματα με τρόπο τίμιο και ειλικρινή και όσον αφορά και τους στόχους που λέει ότι δεν τους πετύχαμε. Και μετά λέει ο εισηγητής ότι δεν υπήρχαν, δεν έγιναν αρκετές ε, διαρθρωτικές ε, μεταρρυθμίσεις, ε, κάτι με το οποίο θα ήθελα να συμφωνήσω. Οι συνάλφοι από την Ιρλανδία και την Κύπρο επίσης μας είπαν ποιες προόδους επέτυχαν μέσω των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και τέθη από κάποιους συναδέλφους το ζήτημα του πώς μπορούμε να βλύνουμε τις ε, ανισότητες. Η απάντηση είναι με το να αμβληθούν ε, οι διαφορές στην ανταγωνιστικότητα των οικονομιών μας. Αυτό δεν είναι απλό και χρειάζονται βεβαίως για αυτό πολιτικές πλειοψηφίες και βεβαίως γι' αυτό υπάρχει αν έχει και πείσει κανείς την πλειοψηφία της κοινωνίας ότι είναι αναγκαίες οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Αυτό είναι πολιτικά πολύ δύσκολο και το γνωρίζουμε πολύ καλά στη Γερμανία. Η έκθεση, ούτως ή άλλως, λέει ότι η Γερμανία πριν από 20 χρόνια ήταν ο μεγάλος ασθενής της Ευρώπης. Ότι ακριβώς λόγω της έλλειψης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων είχε μείνει πίσω. Γι' αυτό οι διαρθρωτικές αυτές μεταρρυθμίσεις στις χώρες μας είναι το κλειδί. Και το ότι ρίχνει εκεί το βάρος ο εισηγητής είναι πάρα πολύ θετικό και μπορούμε να το στήριξουμε. Μια κουβέντα για αυτό το οποίο ακούστηκε το ποια δημοκρατική νομοποίηση έχει το Eurogroup. Θεωρώ πως θα πρέπει να θυμόμαστε ότι οι Υπουργοί Οικονομικών ε, του Eurogroup βεβαίω έχουν δημοκρατική νομιμοποίηση μέσω των Εθνικών Κοινοβουλίων και των πλειοψηφίων που έχουν, των πλειοψηφιών που έχουν στις ε, κοινωνίες τους. Δηλαδή να λέμε ότι δεν έχει δημοκρατική νομιμοποίηση το Eurogroup δεν ισχύει, όλα τα μέλη του έχουν τη δημοκρατική νομιμοποίηση στις χώρες τους. Μία παρατήρηση ακόμα για την Γερμανία. Έχω την τιμή να εκπροσωπώ την ε, Γερμανική Ομοσπονδιακή Συνέλευση. Έχουμε εμείς σε επίπεδο κρατηδίων και ομοσπονδίας το λεγόμενο φρένο χρεών ισχύει για τα κρατήδια από το 2020, κάτι το οποίο έχει μακροπρόθεσμα βεβαίως το αποτέλεσμα ότι θα έχουμε περιθώρια για επενδύσεις. Το βλέπουμε. Η ίδια Ομοσπονδία το 2014 ε, τήρησε το φρένο των χρεών και έτσι αύξησε κατά πολύ τις επενδύσεις γιατί είχε πλέον, ε, έχοντας να εξυπηρετήσει λιγότερα χρέη, περιθώριο για περισσότερες επενδύσεις. Σας ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Περβάνς Μπερές, συντονιστής της Ομάδας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ευχαριστώ πολύ, αξιότιμε Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Είναι πάντα σημαντικό να είμαστε εδώ και να ανταλλάσσουμε απόψεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Το δεύτερο ήμιση του έτους όπου κάνουμε έναν απολογισμό για να δούμε πού βρισκόμαστε εγώ θέλω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις που θεωρώ ότι είναι επίκαιρες ακόμη και για τη σημερινή μας τη συνάντηση. Πρώτα απ' όλα, πέρυσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέσπισε την αρχή του Aggregate Fiscal Stance, του ομαδοποιημένου αυτού του προσανατολισμού. Στο Συμβούλιο και σε ορισμένα κράτη-μέλη αυτό προκάλεσε έντονες συζητήσεις. Αν θέλουμε να έχει συνεκτικότητα αυτό που είναι αναγνωσμένο, ότι δηλαδή το ΕΦΣΥ για να πετύχει θα πρέπει να έχουμε μια μακροοικονομική προσέγγιση με, αυτή τη θετική, με αυτό το θετικό μαδοποιημένο προσανατολισμό για τα δημοσιονομικά. Και με τα εθνικά κοινοβούλια νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε τη μάχη στην πρώτη γραμμή του μετόπου. Η συνάδελφος Κρέτσο από τη Ρουμανία είπε κάτι που θέλω και εγώ να αναφέρω. Ευρωζώνη, μη ευρωζώνη. Είναι μία συζήτηση που μας διχάζει αδίκως, κατά την απόψή μου. Όταν έκανε την ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης ο πρόεδρος Γιούνκερ, πρότεινε την ε, συγκρότηση ενός πρωταξιακού ταμείου, ε, δηλαδή πριν την ένταξη μιας χώρας, πριν την προσχώρησή της στην Ευρωζώνη. Φέρει να αυτά έλεγα εγώ αν ήμουν Αγγλίδα. Αλλά αν θέλουμε ένα τέτοιο ταμείο, τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει σαφής δέσμευση ως προς το χρονοδιάγραμμα της προσχώρησης μιας χώρας στην Ευρωζώνη. Διότι σε διαφορετική περίπτωση τα διαφορετικά ταμεία έχουν το ρόλο τους για τη σύγκληση. Γιατί να τα αντικαταστήσουμε. Αν ο στόχος προσχώρηση στην Ευρωζώνη ξαναπάρει πολιτικό χαρακτήρα και αρχίσει να συζητείται σε πολιτικό επίπεδο και για την Ευρωζώνη και για τα κράτη-μέλη που δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη, αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να το σκεφτούμε και όχι να αρνούμαστε ότι τελικά υπάρχει μια διαφορά. Δεν είναι το ίδιο. Πώς θα το κάνουμε τώρα να είναι κάποιος μέλος της Ευρωζώνης και να μην είναι μέλος της Ευρωζώνης. Δεν μπορούμε να παριστάνουμε ότι είμαστε όλοι στην Ευρωζώνη. Το ζήτημα των επενδύσεων είναι ένα ζήτημα που τίθεται για το σύνολο της Ευρωπαϊκή οικονομίας. Το ίδιο και η οικολογική μετάβαση που αφορά όλη την ευρωπαϊκή οικονομία συνολικά. Δεν μπορούμε όμως να αγνοούμε ότι το πότε η τάδε δίνα χώρα θα μπει στην Ευρωζώνη είναι σημαντικό, είναι κρίσιμο σημείο. Επίσης πρέπει να έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων για το πακέτο που θα θέσει επιτάπητος η Κομισιόν στις 6 Οκτωβρίου. Το έθεσε ουσιαστικά. Και θα πρέπει να βρούμε την ισορροπία και από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το δημοκρατικό ζήτημα της διακυβέρνηση είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά ο πρόεδρος μου κάνει σήματα και δεν μπορώ να αναπτύξω αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Ελπίζω να το κάνουν άλλοι που θα έρθουν μετά από μένα συζήτηση. Φυσικά, περβάς. Και θέλουμε να έχουμε συνεχή διαρκή διάλογο και με τα Εθνικά Κοινοβούλια στο Ταλίν. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση, ελπίζουμε, στη διάσκεψη του Κύριο Σπάλο, Περέιρα, από πού είναι όμως, από το Κοινοβούλιο της Πορτογαλίας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Θα ξεκινήσω από την έκθεση και θα έρθω μετά στα της Πορτογαλίας. Δεν είμαι και τόσο ενθουσιώδης οπαδός αυτής της έκθεσης, διότι, ναι, εντάξει, συμφωνούμε όλοι ότι η ανάπτυξη στο 3% κατά μέσο όρο ε, θα λύσει όλα μας τα προβλήματα να το πετύχουμε αυτό, θα έχουμε ανάπτυξη, θα έχουμε απασχόληση, δημοσιοοικονομικά Το πρόβλημα δεν είναι ο στόχος. Είναι πώς θα τον επιτύχουμε, με τι εργαλεία, με τι μέσα. Η έκθεση περιέργω μα επενθύμησε τι είχε υποθεί στη Λισαβόνα, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2000, ότι σε 10 χρόνια η Ευρώπη θα είναι πιο ανταγωνιστική, δυναμική οικονομία βασισμένη στη γνώση, που θα μπορεί να έχει βιώσιμη ανάπτυξη κτλ. Πάρα πολύ ωραία τα λόγια. Αλλά μας το υπενθύμησε γιατί δεν αρκούν τα λόγια. Χρειάζονται και μέσα, χρειάζονται και εργαλεία. Και αυτά τα εργαλεία και αυτά τα μέσα θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τα εξή προβλήματα. Πρώτον, πώ διορθώνουμε στην Ευρωζώνη τι μακροοικονομικέ ανισορροπίε. Διότι δεν αρκεί να έχει αυτό το μηχανισμό, αυτή τη διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών. Αλλά πρέπει να τι διορθώσει αυτέ τι ανισορροπίε. Έχουμε χώρε όπω η Γερμανία, η Ολλανδία και άλλε χώρε που έχουν υπερβολικό πλεόνασμα. Πώ θα το διορθώσουν. Και ανάποδα, το έλλειμμα επίση. Πώ θα έχουμε αυτή, αυτό τον μέτρο παθώς επεκτατικό δημοσιονομικό προσανατολισμό που είπαν οι στο το είπε ο κύριος Περέρα, ο σκιώτης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχουν λόγοι και ελπίζω να έχω κάποια δευτερόλεπτα για να σα πω γιατί δεν είναι επεκτατικό αυτό ο δημοσιονομικό προσανατολισμό, αυτή η πολιτική στην Ένωση. Γιατί δεν μπορεί να είναι. Πολύ απλά. Και θα σα πω για ποιο λόγο. Τι μέσα θα χρησιμοποιήσουμε στο ευρωπαϊκό επίπεδο για να αυξήσουμε την απασχόληση, για να μειώσουμε την νεανική ανεργία που είναι μεγάλο πρόβλημα. Πρέπει να έχουμε εργαλεία για τις πολιτικέ μας και όχι απλά στόχους. Τώρα, να πω λίγο και για την Πορτογαλία. Η Πορτογαλία έχει πολύ καλό ιστορικό τα τελευταία χρόνια, πολύ καλό ιστορικό επιδόσεων. Δεν έχουμε πλέον το δημοκρατικό έλλειμμα. Είμαστε από το 16 κάτω από το 9% σε ό,τι αφορά το έλλειμμα και τα το χρέο μα ε, είναι γύρω στο 170% κτλ. Αλλά έχουμε τροτά σημεία και έχουμε και μακροοικονομικές ανισορροπίε. Άρα εξακολουθούμε να έχουμε προβλήματα. Δεν βοηθάει και πολύ όμω η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό έχει να κάνει με τη δημοσιονομική πολιτική και είναι και η τελευταία μου σκέψη. Ο μεσοπρόθεσμος στόχο. Όλε έχουμε. Όλε οι χώρες έχουμε μεσοπρόθεσμο στόχο. Για την Πορτογαλία αυτό ο στόχο είναι συν 0,5% Στο ισορροπία το ισοζύγιο. Τι λέει η Ένωση για την Πορτογαλία. Το 2021 θα πρέπει να έχετε πλεόνασμα 4,9%. Ο τρόπος με τον οποίο ορίζεται αυτό το μεσοπρόθεσμο, αυτός ο μεσοπρόθεσμος στόχος ε, για πολλές χώρες ε, απαιτεί ουσιαστικά μια δημοσιονομική πολιτική που δεν είναι καλή για τη χώρα. Στην Πορτογαλία έχουν γίνει μελέτες, μπορώ να σας ε, δώσω τα σχετικά έγγραφα, που δείχνουν ότι με πιο επεκτατική δημοσιονομική πόλη θα έχουμε καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα και χαμηλότερη ε, σχέση χρέους ΑΕΠΑ. Και αυτό ήταν το τελευταίο μου σχόλιο. Ευχαριστώ. από τη Δανία. A ε, micro, micro Tak ευχαριστώ, Πρόεδρε. ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω κυρίως τον κύριο Χέρκμαρκ. Έχει δίκιο ο κύριος Χέρκμαρκ όταν αναφέρθηκε στο κεφάλι στο ψυγείο και τα πόδια στο φούρνο. Έχει απόλυτο δίκιο. Να αναφερθώ όμως και σε κάποια κοινά σημεία στην Ευρώπη και τα οποία θα πρέπει να απασχολήσουν την Κόμισιον και το Κοινοβούλιο. Ξεκινώντας και για τη δική μου χώρα να πω ότι η πολιτική μας η οικονομική θα πρέπει να είναι μια βιώσιμη ουσιαστικά πολιτική. Δυστυχώς η συζήτηση δεν έχει ολοκληρωθεί γύρω από αυτό. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας Στη δική μου χώρα ακόμα και η κυβέρνηση και το κοινοβούλιο τις προκλήσεις αυτές έχει κληθεί πλέον να τις αντιμετωπίσει. Το είδος τώρα ε, της ανάπτυξης ε, πρέπει να εντοπιστεί κυρίως, που παρουσιάζει και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, στον τομέα της ζήτησης. Ορισμένες από τις μεταρρυθμίσεις οι οποίες έχουν εφαρμοστεί και σε μας έχουν τονώσει τις αρνητικές καταστάσεις που βλέπουμε και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Έχουν δηλαδή αρνητικές συνέπειες. Συνεπώς η έλλειψη αυτή ισορροπίας οφείλεται σε λανθασμένες πολιτικές επιλογές. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ακόμα περισσότερους πόρους για την αγορά ομολόγων από τα κράτη-μέλη, από πλευρά της τράπεζας, και θα πρέπει η οικονομία να προσπαθήσει να περάσει στη σχεδίαση νέων προϊόντων που θα την καταστήσουν πιο ανταγωνιστική. Ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών δεν τονώνει την αγορά και δεν τονώνει την οικονομία των κρατών μελών, αλλά τονώνει ουσιαστικά μόνο τις ίδιες τις χρηματοπιστωτικές εταιρείες. Συν της άλλης έχουμε μια οικονομική πολιτική η οποία εξακολουθεί δυστυχώς να σωρεύει χρέη. Έχουμε αυξήσει την, το χρέος μας και σε, στη δική μας περιοχή κατά 57 δις. Συνεπώς λοιπόν η ανάπτυξη της οικονομίας είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να σχεδιαστεί εκ νέου. Και θα πρέπει να δούμε και ποια είναι τα οικονομικά μέσα τα οποία θα έχουμε στη διάθεσή μας. Και εδώ φυσικά η αρχή της ισότητας ελείπει συστηματικά από όλες τις συζητήσεις. Thank you. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαυρίδης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πριν μία εβδομάδα περίπου είχαμε στην Ολομέλεια στο Στρασβούργο μια συζήτηση για το Fiscal Compact, το Δημοσιονομικό Σύμφωνο, και μιλούσαμε για τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών. Θέλω λοιπόν να τονίσω ότι έχουν ήδη αναφερθεί κάποια πράγματα, τα οποία θεωρώ πάρα πολύ σημαντικά. Εάν θα μιλάμε για δημοσιονομικό σύμφωνο, το οποίο να αφορά τη σύγκληση των πραγματικών οικονομιών των κρατών μελών, τότε πρέπει να ξαναδούμε το θέμα και πώς και τι αλλαγές χρειάζονται, ούτω ώστε να έχουμε σύγκληση στις πραγματικές οικονομίες. Εάν κοιτάξουμε από το 2013 μέχρι σήμερα, αντικειμενικά το αποτέλεσμα είναι απογοητευτικό. Τα θέματα που χρήζουν αλλαγών είναι αρκετά και ήδη πολύ σωστά έχουν υποδειχθεί από διάφορους εδώ σε αυτό το δωμάτιο. Για παράδειγμα, εμπλοκή των ιδίων των κρατών μελών στις διαθροτικές τους αλλαγές και όχι επιβολή. One size does not fit all. Ενώ το ξέρουμε, το αναγνωρίζουμε, στην πράξη δεν το εφαρμόζουμε και αγνοούμε τις ιδιαιτερότητες των κρατών μελών. Πρέπει να σεβαστούμε τους κανόνες για διόρθωση μακροοικονομικών ανομαλιών και υπερβολών, αλλά επικεντρώνεται η Κομισιόν περισσότερο στα υπερβολικά ελλείμματα και όχι στα υπερβολικά πλεονάσματα. Θα μπορούσε κάποιος να επιχειρηματολογήσει ότι τα ελλείμματα των μεν είναι εν τα πλεονάσματα των άλλων. Και δύο κουβέντες, έχω ακόμα ένα λεπτό. Do I have one more minute, Chairman? Okay. 45 seconds. Okay, I spend the rest of my 45 seconds on the banking union. When we initially agree on the banking... union, Την Τραπεζική Ένωση λοιπόν. Όταν αρχικά συμφωνήσαμε για την Τραπεζική Ένωση, συμφωνήσαμε για τρεις πυλώνες την διάσωση, τη ρύθμιση και μια πανευρωπαϊκή εγγύηση καταθέσεων. Μετά από τόσα χρόνια, οι δύο πυλώνες έχουν εφαρμοστεί, αλλά ο τρίτος πυλώνας που θα έπρεπε να υπάρχει για να έχουμε ε, ίσους όρους ανταγωνισμού ακόμα εκρεμεί. Πρέπει να το ξαναδούμε αυτό εάν θέλουμε να έχουμε ίσους όρους ανταγωνισμού για όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ Κάρελ Φίτλερ. Από την Βουλή της Τσεχίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βλέπω ότι... Τρία λεπτά δεν είναι ίδια για όλους. Εγώ δες, μαθημένος από το Κοινοβούλιο της Αιχίας σημείωσα κάποια πράγματα. Αρχικά δεν ήθελα να μιλήσω, αλλά ε, τελικά ζήτησα τον λόγο από την συζήτηση. Η συζήτηση μέχρι στιγμής έχει δείξει ότι ε, υπάρχουν τρία χαρακτηριστικά πράγματα. Πρώτα απ' όλα. Υπάρχει ο υποθετικός λόγος που χρησιμοποιούν οι ομιλητές. Τι θα έπρεπε να γίνει, τι θα έπρεπε να έχουμε πετύχει τα λοιπά. Το δεύτερο. Έχουμε τις ε, υποτιθέμενες θετικές προσδοκίες, ε, το λαμπρό μέλλον που μας περιμένει, τις μεγάλες αυτές προσδοκίες για το μέλλον και το τρίτο το οποίο θα να φέρω είναι ότι πολλοί ομιλητές αναφέρουν τις ε, ανισότητες, τις ανισορροπίες, τις απογοητεύσεις, ε, την ατελή νομισματική και δημοσιονομική πολιτική της Ευρωζώνης. Ένας ομιλητής ε, αναφέρθηκε στο ότι δεν υπάρχει μία λύση για όλους, one size does not fit all και συμφωνώ πλήρως. Αυτά τα οποία άκουσα και δεν είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι παρόμοια με αυτά τα οποία άκουσα την προηγούμενη φορά που είχα έρθει εδώ. Και είχα και στο παρελθόν εμπειρίες με το κομμουνιστικό καθεστώς και εκεί πέρα μιλούσαν όλοι για το λαμπρό μέλλον που μας περιμένει, αλλά η πραγματικότητα ήταν διαφορετική. η Ευρώπη πολλών ταχυτήτων ή με την περιφέρεια ή όπως αλλιώς ε, το πούμε, είναι απλά η συνειδητοποίηση του ότι η Ευρώπη δεν λειτουργεί και κάποιοι προσπαθούν να το καλύψουν με ωραία λόγια, με μεγάλα λόγια και λένε Ευρώπη, δύο ταχυτήτων κλπ. Αυτό είναι το βασικό που δεν τολμάει κανείς να πει ε, δημοσίως. Η Ευρώπη πολλών ταχυτών, ταχυτήτων, κατά την άποψή μου, σημαίνει την αποσύνθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Πύρνικ από την ε, ομάδα των φιλελευθέρων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ευχαριστήσω τους συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια που ήρθαν μαζί μας σήμερα να συζητήσουμε ένα τόσο σημαντικό θέμα. Θέλω επίσης και κυρίως να ευχαριστήσω τον κύριο Χέκμαρκ για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε κατά τη διάρκεια των, συζητήσεων για το ε, Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Η έκθεση αυτή είναι μια συμβιβαστική έκθεση. Συνδυάζει τις διαφορετικές θέσεις οι οποίες εξ αρχής υπήρχαν. Ως και όδηση για την ομάδα των φιλελευθέρων θα μου επιτρέψετε να τονίσω το εξή. Επανειλημμένα έχει διευκρινιστεί ότι πάρα πολλέ χώρες δεν έχουν εφαρμόσει τις συστάσεις αυτές και μόνο 2% εφαρμόστησαν πλήρως κατά τη διάρκεια του 2016. Ιδιαίτερα όταν εξετάσει κανείς πιο προσεκτικά τις μεταρρυθμίσεις, εκεί όπου υπάρχει λιγότερη πρόοδος, η εικόνα είναι απογοητευτική. Τα περισσότερα προβλήματα αναφέρονται σε μεταρρυθμίσεις που άπτονται του ανταγωνισμού και της έρευνας και της ανάπτυξης. Αν θέλουμε να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί στο μέλλον και σε αυτούς τους τομείς, όπου θα πρέπει να οδηγεί την κούρσα η Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να αλλάξουμε. Πρέπει να ενισχύσουμε τις προσπάθειες που κάνουμε για την εφαρμογή των συστάσεων αναχώρα η οικονομία ανακάμπτει και στηρίζεται από τις μεταρρυθμίσεις αυτές. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να είναι διαφορετικές. Ο μοναδικός με τον οποίο οι οικονομίες μας θα παραμείνουν ανταγωνιστικές στον σημερινό κόσμο και σήμερα και αύριο είναι η αύξηση της παραγωγικότητας οι ψηλότερες επενδύσεις στην έρευνα θα οδηγήσει σε καινοτομίε, οι οποίες καινοτομίε με τη σειρά του θα δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης και ασφάλεια μακροπρόθεσμα της απασχόλησης. Αυτές ε, δεν θα πρέπει να στηρίζονται οι προσπάθειες και οι επενδύσει από περισσότερα χρήματα, αλλά από διαφορετική χρήση των χρημάτων αυτών. Τα τελευταία χρόνια εμείς ε, κατανοήσαμε τη μεγάλη σημασία που έχει η προσπάθεια η οποία γίνεται. Συνεπώς, θα πρέπει ε, να εδώ επισημάνω και το πρόβλημα που μπορεί να έχει το υψηλό χρέος στην περίπτωση αύξησης των επιτοκίων στο μέλλον. Αυτό θα πρέπει λοιπόν να το λάβουμε υπόψη μας και θα πρέπει ταυτόχρονα να πάρουμε μέτρα για την ενίσχυση των διασυνοριακών μορφών εμπορίου και συνολικά την ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς. Ευχαριστώ. Τελευταίος ομιλητής και θα κάνω και εγώ κάποιες πολύ σύντομες παρατηρήσεις, αλλά πρώτα θα μιλήσει ο κύριος Χέιζ από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε σύντομα να καλωσορίσω τους συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια και ειδικά τον συμπατριώτη μου, τον κύριο Ντόναλ. Το σημαντικότερο θέμα που προκύπτει εδώ είναι η αναγκαιότητα της ιδιοκτησίας, όπως λέγεται, από τα κράτη-μέλη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Δεν θα η Ευρώπη καλύτερο μέρος από πλευράς παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας αν δεν εφαρμοστεί η ατζέντα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Στη χώρα μου θέσαμε στους Ιρλανδούς σε δημοψήφισμα την συνθήκη του Δημοσιονομικού Συμφώνου σε πολύ δύσκολες στιγμές ο κόσμος ε, κάθε γενιάς δεν θέλουν ε, δεν θέλει να ξαναζήσει το γράμμα που είχε με την κατάρρευση των δημοσίων επενδύσεων. Και αυτό το οποίο κάναμε είναι ότι έχουμε τώρα κάποιους κανόνες στο εξαπλό και στο διπλό πακέτο που πρέπει να εφαρμόζονται για όλους, μεγάλους και μικρούς. Αυτό δεν συνέβη στο πρώτο μέρος δεκαετίας του 1990. Οι κανόνες είναι οι ίδιοι για όλους και πρέπει να μείνουμε σε αυτούς ανεξαρτήτως του μεγέθους των κρατομελών. Και τέλος κύριε Πρόεδρε, η σημασία των συστάσεων αναχώρα στο εξάμεινο είναι να καθοδηγούν τα κράτη-μέλη για να κάνουν πράγματα που είναι προς το μακροπρόθεσμο συμφέρον τους. Και αυτό σημαίνει ότι η Κομισιόν δεν πρέπει να κάνει αντιγραφή κάθε χρόνο των ίδιων συστάσεων, αλλά να συνεργάζεται με τα εθνικά κοινοβούλια για να υπάρχουν συστάσεις ε, που θα έχουν αυτή την λεγόμενη ιδιοκτησία. Εμεί σε κάποια φάση είχαμε ένα έλλειμμα 20% του ΑΕΠ και χρειάστηκαν 10 χρόνια να το διορθώσουμε και τώρα θα έχουμε ισοσκελισμένο προϋπολογισμό του χρόνου στο, το 2018. Αυτό είναι παράδειγμα του δύσκολου δρόμου που έπρεπε να ακολουθήσουμε και δεν θα επαναληφθεί εάν τηρήσουμε τους κανόνες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και εγώ. Ποιος άλλος ζήτησε τον λόγο και πάλι. Ναι. Ο κύριος Κράινερ από την Αυστρία. συγγνώμη δεν σας είδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θα έλεγα ότι δεν μου αρέσει η έκθεση στο σύνολό της, αλλά κάποια τμήματα της είναι πολύ ιδεολογικά και δεν μοιάζουν τόσο αντικειμενική περιγραφή της κατάστασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έλεγα ότι ακόμα και νεοκλασικοί οργανισμοί όπως ο ΣΑΡΑ, πλέον σταμάτησαν να γράφουν έτσι πριν από 10 χρόνια. Π.χ. η σύσταση να κοπούν απλά οι δημόσιες δαπάνες και όλα θα πάνε καλύτερα είναι τόσο πολύ πρώτη κρίση και πραγματικά ανησυχώ που δημοσιεύεται κάτι τέτοιο σήμερα. Γνωρίζουμε πως οι χώρες που παραδοσιακά έχουν πολύ υψηλό, μεγάλο δημόσιο τομέα η Σουηδία και Δανία πηγαίνουν πολύ καλά παρά το ότι έχουν μεγάλο και όχι παρά το ότι έχουν δημόσιο τομέα αλλά επειδή έχουν πολύ αποτελεσματικό δημόσιο τομέα. Το θέμα λοιπόν όσον αφορά τον δεν είναι πώς ε, τον περικόπτουμε, αλλά πώς θα γίνει πιο αποτελεσματικός. Και νομίζω ότι αν αντικειμενικά δούμε τις ε, κοινωνίες μας ε, και το πώς λειτουργούν, όχι από ιδεολογική αλλά από ρεαλιστική σκοπιά, θα έλεγα πως οι επενδύσεις, οι δημόσιες μπορεί να είναι και καλύτερες από τις ιδιωτικές. Πρέπει να δούμε λοιπόν πως θα ενισχυθεί ο δημόσιος τομέας και θα γίνει πιο αποτελεσματικός και όχι μόνο να περικοπεί. Ελπίζω η έκθεση να ξαναγραφτεί πριν ψηφιστεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δώσατε τον λόγο. Πριν ε, δώσω το λόγο μου στο ξανά στον Σίδη, θα κάνω και εγώ κάποια σχόλια. Βεβαίω, ευκρινίζοντα ότι έχουμε ένα σχέδιο έκθεσης ε, και ο εισηγητής ε, θα προετοιμάσει κάποιες συμβιβαστικές ε, τροπολογίες. Αυτό το λέω σε αυτούς που θεωρούν ότι δεν είναι ισορροπημένη έκθεση. Βεβαίω είναι μια έκθεση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που εκφράζει κάποιες συγκεκριμένες απόψεις. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε έναν συμβιβασμό. Και ε, δούμε και το ιστορικό των τελευταίων ετών, νομίζω θα βρεθεί κάποιο πεδίο συμβασμού, γιατί είναι να αναγνωρίσουμε γιατί τώρα έχουμε ανάκαμψη, νομίζω ότι θα δούμε ότι αυτό γίνεται ε, χάρη σε πολλά στοιχεία βεβαίως. Οι χώρες εκείνες οι οποίες έκαναν μεταρρυθμίσεις ε, τα πηγαίνουν καλά και έχει μεγάλη σημασία αυτό να γίνουν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Από την άλλη, εάν συγκρίνουμε το τι έγινε τα τελευταία τρία χρόνια. Εάν ε, δηλαδή μπορούμε να αποφύγουμε μια υπερβολικά κυκλική οικονομική εξυγίανση και μείωση του ελλείμματος ε, για να μην φτάσουμε σε μια κατάσταση όπου θα είναι υπερβολικά αυστηρή η μείωση του ελλείμματος και θα ε, σταματήσει την ανάπτυξη. Οπότε μια πιο ισορροπημένη πολιτική νομίζω έχει αποδειχθεί πιο αποτελεσματική από αυτό το οποίο γινόταν το 2011, 12, 13. Και βεβαίως ε, αναγνωρίζεται τώρα ότι υπήρξε μια υπερβολική εξηγένση και είχε κάποια αποτελέσματα που ενίσχυσαν τον οικονομικό κύκλο βεβαίως και αναγνωρίζουμε τον ε, κεντρικό ρόλο της Ευρωπαϊκής ε, Κεντρικής ε, Τράπεζας. Αν δούμε λοιπόν τις τωρινές προκλήσεις μπορούμε να δούμε ότι ούτε το όραμα αυτών που λένε ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις από μόνες τους θα λύσουν τα προβλήματα. Τηρήστε τους κανόνες και τα πράγματα θα πάνε καλά ούτε αυτοί που λένε όχι χρειάζεται μόνο να υπάρξει κάτι στην δημοσιονομική πλευρά, στην πλευρά των ταπανών και δεν χρειάζεται να γίνουν μεταρρυθμίσεις, έχουν δίκιο. Βεβαίως πρέπει να υπάρξει η κατάλληλη πλευρά δημοσιονομική και βεβαίως όταν τα πράγματα πάνε καλά να σφίξουμε λίγο τα λουριά και αντιστρόφως αλλά και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και το τι σημαίνει αυτό ναι, είναι κάτι το πολύ ενδιαφέρον γιατί θεωρώ ότι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις δεν είναι μόνο να μειώνουμε το κόστος αλλά να ενισχύουμε την ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα, την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης και τα λοιπά. Και έτσι ερχόμαστε στο τελευταίο σημείο που ήθελα να πω που σχετίζεται βεβαίως με αυτό το θέμα και αλλά και την ευρύτερη συζήτηση. Το πώς θα έχουμε μια καλύτερη διοίκηση, το πώς θα έχουμε την κατάλληλη δημοσιονομική στάση, το πώς θα δοθεί προτεραιότητα στις επενδύσεις, καλύτερη ποιότητα δημοσίων δάπανων και σύγκληση οικονομικής πολιτικής και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Γιατί, αν δούμε γιατί, το, γιατί τα πήγαμε καλύτερα τα τελευταία χρόνια, νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι μια καλύτερη διοίκηση θα, και διακυβέρνηση θα βοηθούσε την νομισματική μας ένωση. Υπάρχουν βεβαίως διαφορετικές απόψεις από αυτού και η Κομισιόν θα καταθέσει μια πρόταση για την δημοσιονομική ικανότητα της κοινότητας και έχουμε και την συζήτηση στο Ταλίν η οποία πρέπει να συνδεθεί με αυτήν εδώ την συζήτηση και να βρεθεί το κατάλληλο μείγμα πολιτικής στην τωρινή συγκυρία για να έχουμε μία συζήτηση προσανατολισμένη προς το μέλλον για την εμάθηση και την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Ευχαριστώ, Γκούναρ τώρα. Thank you and, uh, thanks for... Σας ευχαριστώ για τις σκέψεις όλων σας. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε μια κομματική πολιτική συζήτηση εδώ τώρα. Είναι σαφές ότι έχουμε διαφορετικές απόψεις στον τομέα της οικονομίας ανάλογα με την πολιτική μας καταγωγή και προέλευση. Θα μου έκανε εντύπωση να μην συνέβαινε κάτι τέτοιο. Έχει σημασία όμως να βλέπει τον τρόπο με τον οποίο εκφράζονται όλες αυτές οι απόψεις και νομίζω ότι τρία πράγματα είναι αυτά τα οποία θα πρέπει να υπογραμμίσουμε. Πρώτον, Οι οικονομικές πολιτικές είναι περίπλοκα πράγματα. Νομισματική πολιτική, φορολογική πολιτική, διαρθρωτικές αλλαγές, ανταγωνιστικότητα, όλα αυτά θα πρέπει να ενταχθούν στα πλαίσια μιας λογικής. Και νομίζω εδώ ότι το πραγματικό πρόβλημα δεν ήταν όταν έχουν ελλείμματα τα κράτη-μέλη, αυτό σε επίπεδο αντικυκλικής, αν θέλετε, λογικής μπορεί να είναι σχετικά χρήσιμο. Το θέμα είναι ότι μακροπρόθεσμα δεν έχει κανείς ε, τις απαιτούμενες πιστώσεις, την απαιτούμενη ρευστότητα. Και αυτό είναι κάτι που βλάπτει όλες τις οικονομίες. Είπε κάποιος από τους συναδέλφους που προηγήθηκαν ότι θα πρέπει να τηρήσουμε τους κανόνες τους οποίους έχουμε θέσει όχι για να μην έχουμε ελλείμματα, όχι μόνο για να κινητοποιήσουμε τις οικονομικές δραστηριότητες, αλλά για να πετύχουμε την ισορροπία την οποία χρειαζόμαστε. Θα συμφωνήσω ότι πολλές φορές κάποια καταστάσεις που δημιουργούνται δεν βοηθούν στην επίτευξη των στόχων αυτών. Αλλά είναι καλό να γνωρίζει κανείς το πού θέλει να βαδίσει. τα άσχημα νέα για όλους μας είναι ότι η ευρωπαϊκή οικονομία δεν πάει τόσο καλά όσο θα έπρεπε. Τα καλά νέα είναι ότι δεν κάνουμε αυτό το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Δεν έχουμε εξαντλήσει τις δυνατότητές μας. Αν τις είχαμε εξαντλήσει η κατάσταση θα ήταν πραγματικά απογοητευτική. Από τη συζήτηση όμως αυτή βγαίνει και το είπαν ξεκάθαρο ορισμένοι συνάδελφοι, το πώς θα υπάρξουν αλλαγές. Κάποιοι από τους συναδέλφους είπαν ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει από την βαριά κρίση, έχει οδηγήσει στην σταθερότητα σε πάρα πολλές χώρες. Αυτό είναι προφανές αλλά λέει και πολλά. Λέει ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι ακόμα περισσότερο. Μιλάμε για μια οικονομική έκθεση. Είναι αυτονόητο όμως ότι όταν μπορούμε να διασφαλίσουμε τις επενδύσεις, ε, τότε θα αναπτυχθεί η οικονομία με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και ένα τελευταίο σημείο είναι η ανάγκη πράγματι οι μεταρρυθμίσεις να θεωρούνται η ιδιοκτησία της κάθε χώρας και ταυτόχρονα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο να κάνουμε αυτά τα οποία μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούμε να πετύχουμε. Ένα από τα προβλήματα το οποίο παραμένει και θα το θέσω απλά, αλλά είναι κάτι το οποίο με προβληματίζει, είναι ότι ακόμα και αν έχουμε μια οικονομική ανάπτυξη, ακόμα και αν βελτιώνεται η ροή των επενδύσεων, είναι πολύ χαμηλά. και μάλιστα σε μια εποχή νομισματικής πολιτικής ακραίας θα έλεγα με μηδέν επιτόκια. Πώς μπορούμε λοιπόν να διασφαλίσουμε περισσότερες επενδύσεις. Ίσως με μέτρα σε επίπεδο φορολογικό, σε επίπεδο δημοσιονομικό. Ίσως και εκεί θα πρέπει να υπάρξουν μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς μας. Σας ευχαριστώ αλλά με αντιμετωπίσατε με τόση καλοσύνη, ιδιαίτερα τα τελευταία λεπτά. Ε, σας ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που έχουμε μαζί μας τα μέλη των κοινοβουλίων, αν το επιθυμούν, και μπορούμε να θέσουμε ορισμένα θέματα όπως ε, οι ε, φορολογικές μεταρρυθμίσεις, και όπως το CCCTB. Θα δώσω το λόγο στον Λούντεκ Μάγια για να παρουσιάσει το δεύτερο τμήμα της ε, κοινή μας ημερήσιας διάταξης. Ευχαριστώ Ρομπέρτο. Θα ήθελα να ξεκινήσω χωρίς ε, καθυστέρηση. Έχουμε δυστυχώς μείνει λίγο πίσω και θα πρέπει να τελειώνουν οι συνεδριάσεις μας έγκαιρα. Το δεύτερο τμήμα λοιπόν έχει σαν στόχο κάποιες ε, ιδιαίτερα σημαντικές προτάσεις. Την κοινή βάση επιβολής λοιπόν φόρου, την πρόταση η οποία γίνεται, το CCCTB, το πακέτο αυτό έχει σαν στόχο την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς και την ε, αντιμετώπιση των ε, επιθετικών προγραμμάτων φορολογίας στις οποίες στοχεύουν οι μεγάλες επιχειρήσεις. Είναι ένας από τους πιο προβληματικούς τομείς του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο. Ξέρετε ότι τα τελευταία χρόνια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασχολήθηκε με τα Panama Leaks, τα Lux Leaks, όπως επίσης και την πρωτοβουλία των πολιεθνικών για την βελτίωση της κατάστασης στον τομέα της φοροαποφυγής στη φορολογία των μεγάλων επιχειρήσεων. Εν πάση περιπτώσει χαίρομαι που συζητάμε το θέμα αυτό σήμερα με τα μέλη των κοινοβουλίων των κρατών μελών. Η προθεσμία ε, επικουρικότητας είναι η 3η Ιανουαρίου και ήδη έχει υπάρξει ο έλεγχος από 19 κοινοβούλια, ε, Σουηδία, Ολλανδία, Λουξεμβούργο έχουν καταθέσει ε, δύο γνωμοδοτήσεις, ε, μία για κάθε σώμα κοινοβουλευτικό. Η ΕΚΟΝ λοιπόν γι' αυτό ακριβώς αποφάσισε να προσκαλέσει όλους τους εκπροσώπους των κοινοβουλίων των κρατών μελών για να συζητήσουν θέματα όπως η φορολογία της ψηφιακής οικονομίας. Γιατί νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει αμοιβαία κατανόηση ανάμεσα σε εμά και εσάς. θα προχωρήσουμε στην παρουσίαση του κυρίου Τάνκ και του κυρίου Λαμασούρ και μετά θα δώσουμε το λόγο στους εκπροσώπους των κοινοβουλίων που το επιθυμούν. Πριν από τη συνάντηση αυτή πήρατε ένα σημείωμα με τα βασικά χαρακτηριστικά της συζήτησης αυτής και οι δύο αυτές προτάσεις είναι περίπλοκες προτάσεις. Και ελπίζω λοιπόν ότι η συνάντηση αυτή παρά το σύντομο χρονικό της πλαίσιο θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τα ωφέλη και την ουσία της πρότασης αυτής. Επαναλαμβάνω ότι η διαδικασία παραμένει όπως ήταν γνωστή, παρακαλώ να είστε σύντομοι. Οι δύο εισηγητές από 7 λεπτά, Τάνκ και Λαμαζούρ, και μετά τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή των Κοινοβουλίων των Κρατών Μελών έχουν την δυνατότητα να θέσουν ορισμένα θέματα μέχρι 3 λεπτά. Θα είμαστε αυστηροί στο χρόνο. Τρία λεπτά. Ο κύριος Τάνκ. Ευχαριστώ και καλωσορίζω και τους συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Το εκτιμώ. Υπάρχουν δύο προτάσεις επί τάπητος ε, και δύο εισηγητές. Ο Αλένα Μασούρ και εγώ αποφασίσαμε εξ αρχής να συνεργαστούμε στενά γιατί θεωρήσαμε ότι είναι ένα το θέμα και ε, αυτό έπρεπε να γίνει από την αρχή. Δηλαδή λέγαμε ότι η διευθέσει είναι ένα θέμα. Εάν ε, χρειάζεται βεβαίως ε, να δούμε την κοινή βάση των, της φορολογίας των εταιριών θα πρέπει να περιλαμβάνει και τις ε, ΜΚΕ και τον τρίτο πυλώνα γενικούς. Είναι πολύ θετικό το ότι βρίσκεστε εδώ. Ο Λέν Λαμασούρ και εγώ προσπαθούμε να έρθουμε σε επαφή με τα εθνικά κοινοβούλια. Ε, το συζητήσαμε εδώ μέσα και βεβαίως ε, συμβουλεύουμε και τις ε, κυβερνήσεις και θέλουμε να έρθουμε σε επαφή μαζί σας για να τεθεί το ζήτημα αλλά να ακούσουμε και τις δικές σας ανησυχίες και να βελτιώσουμε την πρόταση. Γι' αυτό ακριβώς κάναμε κάποιες επισκέψεις σε κοινοβούλια. Δεν μπορέσαμε να επισκεφτούμε και τα 28 κρατημέλη. Ξεκινήσαμε από το Ταλίν, το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο, την Χάγη, Βερολίνο, Παρίσι και Σόφια. Δείξουμε ότι εκτιμούμε την συνεισφορά των Εθνικών Κοινοβουλίων και να λάβουμε υπόψη τις ανησυχίες τους, αλλά και να θέσουμε το θέμα. Γιατί η πρόταση είναι ένα βήμα στον 21ο αιώνα, ένα δυνητικό βήμα. Είναι μια σημαντική αλλαγή στο φορολογικό σύστημα, είναι μεταρρύθμιση, είναι εξυγχρονισμός, γιατί, γιατί το τρέχον σύστημα φορολογίας εταιριών, με ίσως μια εξαίρεση, ε, δεν είναι του 21ου αιώνα. Είναι από μια εποχή που υπήρχαν τσιμινιέρες και εργοστάσια και εργατιά. Και βλέπαμε όπου, πού ήταν το εργοστάσιο και εκεί πέρα ήταν η πηγή του κέρδους. Και αυτό έχει αλλάξει. Λόγω της παγκοσμιοποίησης. Και έτσι οι μεγάλες πολυεθνικές μπορούν να κάνουν φορολογικό σχεδιασμό, να επιλέξουν το που θα έχουν το κεφάλαιο, τις ψηφιακές πλατφόρμες ε, ε, και την πνευματική ιδιοκτησία εκεί, δηλαδή όπου θα έχουν λιγότερους φόρους. Και έχει οδηγήσει σε μια κατάσταση όπου οι μεγάλες πολυεθνικές πληρώνουν λιγότερο από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μάλιστα, αν δούμε ε, την έρευνα σε διάφορες χώρες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, πληρώνουν ε, κατά μέσο όρο ένα τρίτο περισσότερους φόρους από τις πολυεθνικές. Δεν είναι αυτή η σίγουρη του Και πλέον ε, νομίζω πως ο κόσμος το θεωρεί δίκαιο. Το βλέπουμε αυτό σε αντιδράσει για το LuxLeaks και το πάνω Οι μεγάλες επιχειρήσεις να πληρώνουν λιγότερους φόρους από ένα μαγαζάκι, μια καφετέρια ή ένα βιβλιοπωλείο ή από εσάς και εμένα. Λοιπόν, οι δύο αυτές εκθέσεις προσπαθούν να το αλλάξουν αυτό, εστιάζοντας ε, περισσότερο σε απτούς ε, παράγοντες ε, και αποφεύγοντας όλα τα οικοδομήματα αυτά που επιτρέπουν στους πολυεθνικές να κάνουν αυτόν τον φορολογικό σχεδιασμό που ελαχιστοποιεί ε, τους φόρους. Κοιτάω και το χρόνο. Τούτων λεχθέντων λοιπόν, για να θέσουμε το ζήτημα. Πρέπει να βρεθούν και κάποιοι τρόποι για να βελτιωθεί η πρόταση. Και υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο θα ήθελα να επισημάνω. Είναι η φορολογία της ψηφιακής οικονομίας, των ψηφιακών πλατφορμών Google, Facebook, Amazon, Apple. Εταιρείες οι οποίες είναι ψηφιακές δεν έχουν κάποια σαφή παρουσία ηλικοί ε, στην Ευρώπη και έτσι εύκολα σχετικά αποφεύγουν την πληρωμή των φόρων. Γι' αυτό είχαμε και τις υποθέσεις ε, της Κομισιόν κατά της Apple και της Amazon την προηγούμενη εβδομάδα. Έχει λοιπόν ε, να κάνει αυτό με το τρέχον σύστημα φορολογίας των επιχειρήσεων που απαιτεί κάποια μόνιμη εγκατάσταση και αυτό σημαίνει φυσική παρουσία και όχι ψηφιακή παρουσία. Οπότε ο Αλένα Μασούρ και εγώ προσπαθήσαμε να περιλάβουμε την φορολογία της ψηφιακής οικονομίας, να καθορίσουμε την έδρα με τρόπο διαφορετικό περιλαμβάνοντας και την ψηφιακή παρουσία και αλλάζοντας την κλίδα κατανομής για να περιλάβει και την ψηφιακή εκπροσώπηση. Το επισημαίνω αυτό γιατί είδαμε τις τελευταίους μήνες μια πολύ θετική συζήτηση για το πώς θα έπρεπε η Ευρώπη να φορολογήσει αυτές τις ψηφιακές πλατφόρμες όπως το Google και το Facebook. Μία γρήγορη μελέτη που κάναμε δείχνει ότι, για να σας δώσω ένα παράδειγμα, τα τελευταία τρία χρόνια το Facebook και η Google απέφυγαν 5 δισεκατομμύρια σε φόρους στην Ευρώπη. Πολλά λεφτά, ε, σε τρία χρόνια μόλις. Τώρα, ε, βλέπουμε ότι η Γαλλία είχε μία ιδέα θετική, δηλαδή να βασιστεί ο φόρος στον τζίρο. Νομίζω πως ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εγώ και ο Αλένα Μασούρ τουλάχιστον θέλουμε να περιληφθεί αυτό στην κοινή φορολογική βάση των επιχειρήσεων και να ξεκινήσει αυτό για τις ψηφιακές εταιρείες. Θα μείνω σε αυτά στην εισαγωγή μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε, ε, Πολ, που συνοψίσατε τα βασικά σημεία της πρότασης. Τώρα δίνω τον λόγο στον Αλέν, ο οποίος θα μας μιλήσει για το δεύτερο μέρος στην ενοποιημένη βάση φορολογίας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω από δική μου πλευράς επίσης να σας εκφράσω τη μεγάλη ικανοποίησή μου που είμαι εδώ στην κοινή αυτή συνεδρίαση με τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων. Πριν από κάποια χρόνια ακόμη ήμουν και εγώ μέλος της Γαλλικής Αθηνοσυνέλευσης. Έχω διατελέσει και υπουργό Οικονομικών στη Γαλλία, οπότε αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία στην άποψη των Εθνικών Κοινοβουλίων, ιδίως για αυτά τα ζητήματα που άπτονται της φορολογίας. Και θα ξεκινήσω από το εξή. Σε ό,τι αφορά τα φορολογικά ζητήματα, δεν υπάρχει περίπτωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, παρέμβει σε ζητήματα που είναι εθνική αρμοδιότητα και να θέσει υπό αμφισβήτηση τη φορολογική εθνική κυριαρχία. Οι προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τον οποίο εμεί θα γνωμοδοτήσουμε με την έκθεσή μας, συνάδουν με τι διατάξει της συνθήκη. Και οι αποφάσει λαμβάνονται μόνο με ομοφωνία των κρατών μελών και έπειτα με την έγκριση των Εθνικών Κοινοβουλίων. Άρα τον τελευταίο λόγο τον έχετε εσεί, τα Εθνικά Κοινοβούλια. Έτσι προβλέπουν οι συνθήκε. Όπω είπε και ο Πολ Τάγκ, έχουμε εδώ δύο προβλήματα τα οποία ανέκυψαν λόγω της δημοσιονομικής κρίσης που ξέσπασε πριν από κάμια δεκάρια χρόνια αλλά και από τα σκάνδαλα του τύπου LuxLeaks που ξέσπασαν πριν απο τρια τρία-τεσσέρα χρόνια. Και όλα αυτά έδειξαν τα εξή. Πρώτον, ότι κάποιες πολυεθνικές επιχειρήσεις ε, στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης, κάποιες πολυεθνικές λοιπόν που δραστηριοποιούνται στις πέντε υπήρους, ε, αξιοποιούσαν όλες τις δυνατότητες που τους προσέφεραν οι διαφορετικές φορολογικές νομοθεσίες των κρατών μελών για να φοροαποφύγουν για να αποφύγουν μεγάλο μέρος των φορολογικών τους υποχρεώσεων. Είπε ο Πολ ότι τα φορολογικά συστήματα είχαν σχεδιαστεί για τον 20ο αιώνα, υπήρχαν τότε εξαγωγές σε όλο τον κόσμο, αλλά μια επιχείρηση που παρήγαγε για όλο τον κόσμο, αυτό το έκανε από την χώρα προέλευσης και εξήγαγε στη συνέχεια. Εδώ τώρα έχει ε, υπάρξει εξέλιξη. Αυτές οι αλυσίδες ε, παραγωγής και διανομής ε, καλύπτουν τις πέντε υπήρους. Ένα δεύτερο στοιχείο που ανέδειξαν τα σκάνδαλα και η κρίση είναι ότι και στην ευρωπαϊκή οικογένεια, σε ό,τι αφορά τη φορολογία των επιχειρήσεων, υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών Όχι ότι αυτό είναι κακό, να υπάρχει ένα ανταγωνισμό φορολογικό, εφόσον βέβαια υπάρχει καλή σχέση ε, τιμή εντό και ποιότητα των φορολογικών υπηρεσιών και εφόσον υπάρχουν και τα απαραίτητα φορολογικά έσοδα. Αυτός ο ανταγωνισμός όμως γινόταν αντίθετα με αδιαφανή τρόπο, με αθέμητο και μη δίκαιο τρόπο. Και με βάση αυτά συναγάγαμε, και όταν λέω συναγάγαμε ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή Κομισιόν, Κοινοβούλιο και σε παγκόσμιο επίπεδο ο ΩΣΑ, που όπω ξέρετε δραστηριοποιείται ενεργά στον τομέα αυτό. Συναγάγαμε λοιπόν στο ότι, το ότι χρειάζεται ένα κώδικα δεοντολογία καλή συμπεριφορά σε παγκόσμιο επίπεδο και αυτό ε, προωθεί ο ΩΣΑ με το δικό του σχέδιο δράσης, το οποίο και εμείς έχουμε μεταφέρει στο κοινοτικό δίκαιο με τις ε, οδηγίες μας και σε επίπεδο ευρωπαϊκής οικογένειας αυτό που εμείς πρέπει να κάνουμε είναι να προσαρμόσουμε τα συστήματα φορολόγησης των επιχειρήσεων κατά τρόπο ώστε να παραμείνει η αρχή του φορολογικού ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών Αφενός, αφετέρου όμως, ε, η φιλοσοφία, οι αρχές και οι κανόνες του ανταγωνισμού που εφαρμόζουμε σε όλους τους άλλους τομείς ε, της Ένωσης να ισχύουν και για τα φορολογικά ζητήματα. Δηλαδή να είναι διαφανής ο ανταγωνισμός αυτός, να είναι θεμητός, δίκαιος και αυτό βέβαια περνά αγκαστικά μέσα από την ε, καθιέρωση ενός ενιαίου ορισμού για τα φορολογητέα κέρδη όταν θα καταλήξουμε σε αυτόν τον κοινό ορισμό θα μπορούμε πλέον να καταλήξουμε με πλήρη διαφάνεια και σε κάποιες διατάξεις ό,τι αφορά τους φορολογικούς συντελεστές και, τον... και κάποιους άλλους ορισμούς. Υπάρχει πολιτική συζήτηση. Αν χρειάζεται ένας κατώτης συντελεστής κτλ. Αυτό είναι υποσυζήτηση. Αλλά αυτή είναι η γενική φιλοσοφία. Αυτό που θέλουμε να προσθέσουμε, το είπε και ο Πολ Τάγκ, είναι ειδικέ διατάξεις για την ψηφιακή οικονομία. Με ικανοποίηση διαπιστώνουμε ότι ορισμένες κυβερνήσεις όπως ε, η γερμανική που υπέβαλε σε μια συνεδρία στους G20 τη συνεδρία του Ιουνίου ε, κάποιες σχετικές προτάσει και πιο πρόσφατα Γαλλία θέλουν να δώσουν έμφαση σε αυτό το τομέα και είναι και προτεραιότητα της Αστωνικής Προεδρίας. Σε ό,τι αφορά το ψηφιακό, το ψηφιακό τομέα, δεν θέλουμε μια ειδική προσέγγιση με έναν ειδικό φόρο που θα αφορά μόνο τις ψηφιακές πλατφόρμες. Απλά αυτό που θέλουμε είναι σε ένα κείμενο γενικό για τη φορολογία των πολυεθνικών να μπει και ένα κριτήριο τζίρος για τα ψηφιακά ψηφιακό τζίρο εντό εισαγωγικών. Δηλαδή για να δούμε τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται και είναι αντικείμενο εκμετάλλευση σε ένα κράτο μέλο και αν υπάρχει αυτή η ψηφιακή δραστηριότητα, μια επιχείρηση θα μπορούσε να υπαχθεί στη φορολόγηση των κερδών τη ε, στο κράτο μέλο στο οποίο δραστηριοποιείται. Και βέβαια υπάρχουν και τα ζητήματα του επιμερισμού, της κατανομής. Έχουμε τα κριτήρια που είναι το ενεργητικό, οι πωλήσει και το προσωπικό. Και εκεί προσθέτουμε και τα στοιχεία τα οποία συλλέγονται και είναι μετά σε αυτά τα κράτη-μέλη. Δεν είναι και τόσο θετικά κάποια κράτη. Είναι επιφυλακτικά όχι προς την αρχή, αλλά προς την ιδέα ότι θα μπορούσαν να χάσουν φορολογικά έσοδα εν τέλει. Και φυσικά θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί Άρα θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε κάτι που δεν γίνεται αυτή τη στιγμή, δεν το έχουμε. Μια μελέτη αντικτύπου για να δούμε για τι μεγάλε κατηγορίε επιχειρήσεων, αλλά για όλε τι χώρε επίση. Ποιε θα ήταν οι επιπτώσει ό,τι αφορά τα φορολογικά έσοδα σε σχέση με το προηγούμενο σύστημα. Και το δεύτερο που θα πρέπει να κάνουμε και που προτείνουμε είναι να δημιουργηθεί ένα ταμείο αποζημίωση αντιστάθμισης, ότε τουλάχιστον για μία μεταβατική περίοδο χάρη στην περιστέμενη αξία που θα μπορούσε να φέρει ε, σε κάποιες χώρες, βέβαια θα υπάρξει πρόβλημα για κάποιους άλλους, κάποιο να αντισταθμίζεται αυτόματα, να συμψηφίζεται. Αυτό μπορούμε να τα συζητήσουμε όμως ακόμα. Αυτά είχα να πω, σας ευχαριστώ, Πρόεδρος. Εντάξει, πήρε 30 δευτερόλεπτα από τον Πόλα, αλλά συνεργάζεται πολύ καλά, οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα. Να στραφώ τώρα στους ε, προσκεκλημένους μας από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Ο κ. Σοντών, τρία λεπτά, ο πρώτος ομιλητής από την Ιρλανδία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εμείς θεωρούμε ότι η συζήτηση αυτή παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο κρίσιμο χαρακτήρα θα ζητήσω από τον κύριο Τάν και τον κύριο Ραμασόβ να μας επισκεφθούν στην Ιρλανδία γιατί δεν το έχουν κάνει ακόμα. Εγώ είμαι μέλος της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου. Είμαστε φυσικά μια πολυκομματική επιτροπή. Εμείς έχουμε καταθέσει ακριβώς την πρότασή μας για την πρόταση για το CCTB. Θεωρούμε ότι η πρόταση αυτή παραβιάζει εν πολύ στις δυνατότητες τις οποίες έχουμε σαν κρατομέλος για τον καθορισμό της φορολογικής μας πολιτικής. Αυτό το 12,5% που έχουμε εμείς είναι ένα επίπεδο διαφανέστατο, είναι χαρακτηριστικό συστατικό της οικονομικής μας πολιτικής, είναι κάτι το οποίο θα έλεγα έχει βοηθήσει στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και λειτουργεί καλά εδώ και αρκετά χρόνια και νομίζω ότι το πραγματικό ποσοστό και το θεωρητικό ποσοστό είναι πάρα πολύ κοντά. Η, το σημερινή πρόταση, η σημερινή συγγνώμη, πρόταση λοιπόν για το CCCTB παραβιάζει αν πολύ στις δυνατότητες αυτές που τις οποίες έχουμε. Οι υπολογισμοί οι οποίοι γίνονται και τα στοιχεία είναι αρκετά αυθαίρετα που χρησιμοποιούνται και είναι κάτι το οποίο θα δημιουργήσει προβλήματα σε σχέση με τη φορολογική βάση και την χρήση της φορολογικής βάσης στην Ιρλανδία. Τώρα σε σχέση επίσης και με την πρόταση BEPS του ΟΣΑ. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα έλεγα δεν γίνεται σεβαστό με την πρόταση αυτή. Ο κύριος Λαμασούρα αναφέρθηκε βέβαια στη μελέτη BEPS. είναι κάτι το οποίο μπορεί να ισχύει σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά ταυτόχρονα σε σχέση με τη μεταφορά των τιμών είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη σε όλες, όλη την πραγματικότητα την ευρωπαϊκή. Είμαι και μέλος της Επιτροπής Οικονομικών λοιπόν της, του Κοινοβουλίου μας Έχουμε θέσει τις προτάσεις αυτές ε, υπό εξέταση, τις έχουμε αντιμετωπίσει σοβαρά. Ο κύριος Λαμασούρ, σαν παράδειγμα, αναφέρθηκε στις επιπτώσεις που θα μπορούσε να γίνει με την εφαρμογή της πρότασης αυτής για το CCTB. Μια προκατακτική εξέταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, είπε ότι είναι 0,47% του ΑΕΠ της χώρας δεν νομίζω. Νομίζω ότι εμείς που είμαστε μια μικρή εξαγωγική οικονομία, το ποσοστό το οποίο θα μας στήξει η εφαρμογή των προτάσεων αυτών είναι πολύ υψηλότερο. Οι συντηρητικές εκτιμήσεις δείχνουν ότι θα μπορούσαμε να χάσουμε το 15% ε, του ε, φόρου που μπορούμε να εισπράξουμε σε αιτήσια βάση, δηλαδή 5 ε, σχεδόν δις. Συνεπώς λοιπόν το συγκεκριμένο μέτρο αυτό είναι, έχει βέβαια το πλεονέκτημα να θέτει το πρόβλημα, να θέτει ε, την συζήτηση για το πώς λειτουργούν οι φορολογικές πολιτικές. Αλλά θυμίζω ότι στην Ιρλανδία έχουμε περάσει α, ε, αρκετές ε, διαβουλεύσεις γύρω από τα θέματα αυτά και νομίζω ότι η πολιτική την οποία ακολουθούμε στη χώρα μου είναι αυτή που πρέπει να συνεχίσουμε να ακολουθούμε και συμφωνούν και οι συνάδελφοι. Ε, δεν αναφέρομαι στην ουσία αυτών που είπατε, παρακαλώ αναφέρομαι στο τρίλεπτο, γιατί αλλιώς δεν θα μιλήσουν όλοι. Εμείς δεν θέλουμε να εναρμονίσουμε τίποτα με την πρόταση αυτή, αλλά αυτά θα σας τα πούνε οι δύο εισηγητές, συγγνώμη. Ο κύριος Βότσης τώρα έχει το λόγο από την Κύπρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω με κάποια σχόλια επί, της, επί των προτάσεων και θα καταλήξω με τη θέση της Κυπριακής Βουλής γιατί το θέμα αυτό έχει απασχολήσει και Επιτροπή της Βουλής αλλά και την Ολομέλεια και έχουμε καταθέσει την άποψή μας με γνώμη επί των δύο προτάσεων. Να πω ξεκινώντα ότι οι κανόνε για τον υπολογισμό τη φορολογική βάση μαζί με το φορολογικό συντελεστή επηρεάζουν τα φορολογικά έσοδα και άρα πιθανή αρνητική διακύμαση των φορολογικών εσόδων θα επηρεάσει αρνητικά δημοσιονομικά έσοδα που προορίζονται να χρησιμοποιούν για άλλε προτεραιότητε του κράτου μέλου, ω παραδείγματο χάρη μέτρα κοινωνική στήριξη. Η δικαιοσύνη εντό εισαγωγικών Ενό φορολογικού συστήματο, αφορά κατεξοχήν τα ίδια τα κρατημέλη τα οποία είναι υπόλογα στου πολίτε του. Η CCTB δεν λαμβάνει υπόψη τα επιμέρου πλεονεκτήματα και αδυναμίε τη οικονομική θέση κάθε κράτου μέλους ξεχωριστά και δεν αντιστοιχεί στι τρέχουσε και μελλοντικέ ανάγκε του. Η έκθεση ανάλυση του αντικτύπου που εκπώνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει συνολικά θετικά αποτελέσματα στις επενδύσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση στην ολότητά της. Ωστόσο, δεν έχει αξιολογηθεί κατά τρόπο ασφαλή η έκταση του αρνητικού επηρεασμού των επενδύσεων ξεχωριστά για τα κράτη-μέλη, ειδικά για μικρέ οικονομίε όπω τη Κύπρου, ακούσαμε προηγουμένω και για την Ιρλανδία, για τι οποίε τίθεται και ζήτημα κόστου συμμόρφωση σε ανθρώπινου και οικονομικού πόρου. Περαιτέρω, το διοικητικό κόστο για την περίπτωση εφαρμογή μόνο τη πρόταση CCTB δεν έχει επιμετρηθεί. Το ζήτημα της, φο... της φοροαποφυγής αποτελεί αντικείμενο ρύθμισης τόσο στο πλαίσιο του ΩΣΑ, με το BEPS που αναφέρθηκε προηγουμένως σχέδιο δράσης, όσο και στο πλαίσιο της οδηγίας 2016-1164 Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πάταξη της φοροδιαφυγής, την Anti-Tax Avoidance Directive, την ATAT. Αφότερα τα μέτρα βρίσκονται στο στάδιο της εφαρμογή από τα κράτη-μέλη και δεν υφίσταται οποιαδήποτε ένδειξη ότι τα προαναφερθέντα μέτρα δεν επαρκούν. Από το πιο πάνω και την έκθεση ανάλυσης αντικτύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκύπτει ότι δεν έχουν αιτιολογηθεί επαρκώς τα σαφή πλεονεκτήματα τη ανάληψη δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο με βάση την αρχή της επικουρικότητας. Η πρόταση CCTB εδέχεται να διαταράξει την ισορροπία που επιτεύχθηκε από τι διμερεί συμφωνίε αποφυγή διπλή φορολογία που έχουν συναυθεί μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών, καθώ καθώς κατά σύναψη των συμφωνιών αυτών δεν λήφθησαν υπόψη οι πρόνοιε μια ενδεχόμενη CCTB. Το άρθρο 115 τη συνθήκη για τη Λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που σχετίζεται με την εύρυθμη λειτουργία τη εσωτερική αγορά, εσφαλμένα αποτελεί την νομική βάση για την εκπόνηση οδηγιών για κοινή, φορολογική, για κοινή βάση φορολογία εταιρεών και θα αποτελέσει δικό προηγούμενο αν χρησιμοποιηθεί για αυτή την περίπτωση. Κλείνοντα, εκφράζουμε την απορία μα σε σχέση με την αναγκαιότητα υιοθέτηση των δύο προτάσεων οδηγιών εν ώψη των εισηγήσεων σεναρίων που διατυπώνονται στη Λευκή Βίβλο για το μέλλον της Ευρώπης που εκπώνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και μόνο η ύπαρξη αυτών των εναλλακτικών σενάριων δείχνει ότι δεν υπάρχει επιτακτική ανάγκη για άμεση λήψη τέτοιων μέτρων. Υπό το των πιο πάνω, εκφράζουμε την πλήρη διαφωνία μας με τα λόγω μέτρα. Thank you very much. Now the first speaker from uh, European Parliament, uh, Mr. Vieri. Από το Κοινοβούλιο, κύριος, ε, η κυρία. Από το Κοινοβούλιο ποιος είναι? Είναι πολλές από τις προτάσεις επικοδομητικές και θα βελτιώσουν το κείμενο, ιδίως αυτές που αφορούν ε, την περίληψη των ε, ψηφιακών δραστηριοτήτων. Το θέμα είναι βέβαια να είναι συμβατό αυτό με τις προτάσεις μας. Ε, υπάρχουν κάποιες άλλες αλλαγές που θα επηρεάσουν τη φόρμουλα, τον τύπο και είναι καλό ε, να γίνουν τέτοιε τροποποιήσει για να είναι εξασφαλισμένα τα φορολογικά έσοδα για τα κρατη μελη Δεν είναι τέλεια πρόταση, θα πρέπει να έχουμε υπόψη όμω ε, ότι μπορεί να είναι πολλά τα ωφέλη για τι επιχειρήσει ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα υπάρξει ιδιαίτερο διοικητικό άχθος, γιατί θα μειωθεί κατά πολύ μεγάλο βαθμό το βάρος των των επιχειρήσεων που έχουν αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσουν 28 διαφορετικές διοικήσεις. Και δεν επιτρέπει ε, σε αυτές τις επιχειρήσεις να απολαμβάνουν των ωφελημάτων της ε, νέας αγοράς. Επίσης, θα πλησιάσουμε το πεδίο ανταγωνισμού, ε, το ισότιμο, με τις πολυεθνικές. Κάτι που πάντοτε ήταν στόχος μας. Και τελικός στόχος βέβαια θα πρέπει να είναι να τονώσουμε τον ανταγωνισμό με βάση τους φορολογικούς συντελεστές και τις υποδομές. Αυτό θα κάνει ακόμα πιο ελκυστική την Ευρώπη στις, ε, στους επενδυτές και θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας τέλος. Παρότι δεν μπορούμε να δρούμε με γνώμονα το φόβο για αυτό το νέο σύστημα, θα πρέπει να βάλουμε τα απαραίτητα χέγγια, τι ασφαλιστικέ για να μην έχουμε παρενέργειε και για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε περίπτωση που έχουμε κάποια ανεπιθύμητη συνέπεια ή επίπτωση. Μια από τι απαιτούμενε αλλαγέ, κατά την άποψή μα, είναι και τα δύο συστήματα να τεθούν σε εφαρμογή παράλληλα. Καταλαβαίνω βέβαια ότι εξακολουθούν πολλοί να έχουν τι αμφιβολίε του και γι' αυτό προσωπικά Ζητώ την συμπερίληψη ενό μηχανισμού επίλυση διαφορών ε, για να επιλύει τέτοιε διαφορέ και να προασπίζει τα συμφέροντα όλων από τη στιγμή που οι δύο αυτέ βάσει γίνουν πραγματικότητα. Ευχαριστώ. Thank you very much again as stating the deadline for amendments. ευχαριστώ. Η υπεύθυνη για τροπολογίε έχει ήδη περάσει. Κατατέθηκαν τροπολογίες ε, το τέλος του Σεπτεμβρίου. Κατόπιν ο κύριος από την Πολωνία. Μέχρι τρία λεπτά έχετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, η Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Η πολωνική κυβέρνηση στηρίζει τις ε, δράσεις αυτές σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να διασφαλιστεί ότι τα κέρδη που δημιουργούν οι επιχειρηματικές δραστηριότητες θα πρέπει να φορολογούνται στη χώρα όπου δημιουργούνται. Θεωρούμε ότι έτσι θα μπορέσουν όλες οι χώρες να προχωρήσουν. Υπάρχουν κάποια θετικά αλλά και κάποια αρνητικά στην πρόταση. Πρώτα απ' όλα βεβαίως ε, αυτός ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Μόνο ένα κράτο όμως μπορεί να αποφασίσει το ύψος φορολογίας και τον πιθανό φόρο και την ε, φορολογική βάση. Όταν μιλάμε κατόπιν για την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας επιχειρήσεων έχουμε κάποιες επιφυλάξει για τον διασυνοριακό ορισμό για πιθανές απώλειες. Το τρίτο πιθανό πρόβλημα αφορά ε, τις ε, ειδικέ ε, εκπτώσεις από τον φόρο που αφορούν το ύψος των ιδίων κεφαλαίων της ε, κάθε εταιρεία. Και μετά θα πρέπει να προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε ότι τέτοιες λύσεις δεν θα διαταράξουν τα δημόσια οικονομικά γιατί αυτή τη στιγμή ενοποιηθεί η βάση και μετά μοιραστεί με βάση ένα συγκεκριμένο τύπο ίσως ανακύψουν προβλήματα. Και η πέμπτη επιφύλαξή μας ε, στην πρόταση της Κομισιόν. Η Κομισιόν λέει ότι θα ήθελε να μεταφερθούν κάποιες αρμοδιότητες, να μιλάμε για τοπικά διοικητικά δικαστήρια στο ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί πλέον δεν θα έχει τόσο μεγάλη σημασία το που ε, δημιουργείται η κερδοφορία και η τελευταία μας ε, ανησυχία για τις δύο προτάσεις ε, αφορά την συμμόρφωση με την αρχή της επικουρικότητας. Θεωρούμε ότι τα κράτη-μέλη έχουν ε, την δυνατότητα να απαλείψουν ορισμένες αρνητικές πτυχές της φορολογικής δημοσιονομικής πολιτικής μέσω εθνικών μέτρων. υπήρχε ένας νόμος, πέρασε τώρα 12 Ιουλίου στην Πολωνία, στόχος του οποίου ήταν ε, ακριβώς αυτό. Δηλαδή να μην δημιουργηθούν προβλήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο από την διαδικασία αυτήν. Θεωρούμε επίσης πως η πλειοψηφία των κρατών μελών δεν ε, έχουν κάνει εσωτερικές αναλύσεις και πρέπει να γίνουν αυτές για να ξέρουμε περισσότερες λεπτομέρειες για να μην έχουμε άλλα προβλήματα. Και Πέτερ, θεωρώ ότι όταν ολοκληρωθεί το έργο, ο νέος κανονισμός θα είναι υποφελής για τις επιχειρήσεις και τα κράτη. Σας ευχαριστώ, Φίλερ, για τρία λεπτά και πάλι. Η πρωτοβουλία αυτή για την κοινή φάση φορολογίας επιχειρήσεων και την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας επιχειρήσεων είναι δουλειά της Γαλλίας και της Γερμανίας που προσπαθούν να προστατεύσουν τις αγορές τους που είναι αναποτελεσματικές, μη ελαστικές και άρα λιγότερο ανταγωνιστικές. Η μεθοδολογία υπολογισμού της ε, κοινή ενοποιημένη φορολογικής βάσης ε, πηγαίνει αντίθετα προς τα συμφέροντα των οικονομιών που αναπτύσσονται όπως η Τσεχία. Δεν μπορεί να αλλάξει η μεθοδολογία υπολογισμού της φορολογίας χωρίς ε, να συμφωνήσουν οι χώρες, κάτι το οποίο βεβαίως θα είναι προς το συμφέρον των μεγάλων γαλλικών και γερμανικών εταιριών. Επιτούμε λοιπόν να σταματήσουν αυτές οι διαπραγματεύσεις ε, και το και να γίνει ένα δημοψήφισμα για το εάν οι χώρες θέλουν να παραμείνουν στην Ένωση σε όλες τις χώρες και μόνο τότε να σκεφτούμε νέες πρωτοβουλίες. Ίσως ε, έτσι δεν θα πρέπει να επαναληφθεί η κατάσταση ε, κατά την οποία ξεγέλασαν οι πολιτικοί τον κόσμο εισάγοντας ε, νέες αρμοδιότητες μέσω της συνθήκης της Λισαβόνας. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία στην Τσεχία και εγώ είμαι υποψήφιος ε, ενό εκ των κομμάτων που θα κατέβουν στις εκλογές της ε, Τσεχίας και ο κόσμος θα έχει το δικαίωμα να αποφασίσει. Και ελπίζουμε ότι θα στείλουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση εκεί που ανήκει στο χρονοτούλαπο της ιστορίας ως αποτυχημένο πείραμα. Και μια τελευταία κουβέντα για την κοινή βάση φορολογίων επιχειρήσεων. Ακούστηκε κάτι που θα ήθελα να το επαναλάβω. Δεν υπάρχει ένα μέτρο για όλους. Ένα one size fits all. Σας ευχαριστώ. Now, uh, uh, Fabio De Masi, uh... Φάβιο Ντεμάζη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την ΚΟΕ για τρία λεπτά. Σας ευχαριστώ. Ε, είμαι για δύο εβδομάδες ακόμα ευρωβουλευτής ε, πριν πάω στο Γερμανικό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα έξι λεπτά, αλλά βλέπω δεν γίνεται. Λοιπόν, να πω ότι συμφωνώ με τον Πολ και τον Αλέν ότι το φορολογικό μας σύστημα πλέον δεν ανταποκρίνεται στον σκοπό του. 60% του εμπορίου γίνεται... Ε, εντός ε, των επιχειρήσεων, δηλαδή μιλάμε για ενδομιλικές ε, συναλλαγές ε, και αυτό η φοροαποφυγή δεν αντιμετωπίζεται κοιτώντας μόνο το transfer pricing και το πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων. Όμως η εναρμόνιση της φορολογικής βάσης δεν είναι αυτός ο σκοπός. Για μένα λοιπόν το μέτρο είναι αν οι πολυεθνικές όπως η Apple και η Google θα πληρώσουν περισσότερα μετά από αυτή την πρόταση. Και εδώ πέρα έχω κάποιες ανησυχίες που θα ήθελα να τονίσω. Πρώτα απ' όλα μπορούμε να εναρμονίσουμε τη φορολογική βάση, αλλά αν δεν υπάρχει κάποια ελάχιστη κοινή εταιρική φορολογία, τότε θα έχουμε ακόμη πιο έντονο ανταγωνισμό μέσω του ύψους ε, της φορολογίας. Δεύτερον. Μπορούμε να δούμε αν θα είναι ευρύτερη ή κάπως πιο περιορισμένη η φορολογική βάση. Και εδώ πέρα βλέπουμε πως η Κομισιόν θέλει να επιτρέψει την αναγνώριση διασυνοριακών ζημιών. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κάποια κράτη-μέλη, και το ακούσαμε σήμερα το πρωί, να είναι κατά του της ε, ενοποιημένης ε, βάσης ε, φορολογίας επιχειρήσεων και έτσι δεν θα κοιτάμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ποια είναι τα κέρδη και πώς κατανέμονται μετά στα κράτη-μέλη. Μετά έχουμε την οδηγία για την φοροαποφυγή, κάτι το οποίο εγώ πάντα θεωρούσα ότι είναι το μίνιμουμ. Και κάποια κράτη-μέλη τα οποία είναι πιο φιλόδοξα μπορούν να προχωρήσουν παραπέρα. Τώρα στην πρόταση αυτή βλέπουμε ότι η οδηγία περί θα γίνει το maximum, κάτι που είναι πρόβλημα, γιατί χρειαζόμαστε και μέτρα όπως η φορολογία στην πηγή στο εθνικό επίπεδο για να αντιμετωπίσουμε τις φορολογικές πρακτικές κρατών μελών που δεν είναι διατεθειμένα να συνεργαστούν σε διεθνές επίπεδο. Τρίτον, έχουμε διαφορετικά λογιστικά πρότυπα και εάν έχουμε κοινή βάση φορολογίας επιχειρήσεων αλλά διαφορετικά λογιστικά πρότυπα πρόκειται για ένα τεράστιο δώρο στις ε, λογιστικές εταιρείε, PwC κτλ. Τέταρτον, έχουμε την έκπτωση αυτή της έρευνας και της ανάπτυξης που υπάρχει στο άρθρο 9 και φοβόμαστε ότι αυτή η φορολογία παρόμοια με τα patent boxes δεν θα έχει τελικά θετικό αντίκτυπο στην έρευνα και ανάπτυξη, απλά θα αποτελέσει ε, μεγαλύτερη δυνατότητα για ε, έκπτωση από τον φόρο και δεν πρέπει να το επιτρέψουμε γιατί ήδη υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια για τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε πολιτικές λιτότητε και πρέπει ο κόσμος να εμπιστευτεί ξανά το, Ευρωπα... το έργο της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωση. Ε, ζητήστε τα τρία λεπτά στο Βερολίνο. Λοιπόν, από την Ρουμανία κατόπιν, ο κ. Σοπέα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε να κάνουμε με ένα αντικείμενο το οποίο αφορά στα κράτη-μέλη κυρίως. Εμείς είμαστε υπέρ της αντιμετώπισης του συγκεκριμένου θέματος αυτού σε δύο στάδια. Άλλωστε και οι δύο αυτές προτάσεις πρέπει να αντιμετωπιστούν σαν λύση για να υπάρξει επιτέλους ένα δίκαιο σύστημα φορολογίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συν της άλλης ε, θα έλεγα η κυριαρχία της ψηφιακής οικονομίας είναι κάτι το οποίο αφορά σε όλες τις χώρες μέλη και είναι κάτι το οποίο, στο οποίο θα πρέπει να βρούμε μία λύση. Η δεύτερη φάση του CCTB μας απασχολεί βέβαια γιατί επηρεάζει κατά κάποιο τρόπο ε, τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Στόχος αυτών των ρυθμίσεων είναι να φορολογείται το κέρθος εκεί όπου παράγεται. Γι' αυτό κύριε Λαμασούρ πώς ακριβώς βλέπετε τη λειτουργία του Ταμείου Αντιστάθμισης. Θα απαντήσει ο κύριος Λαμασούρ στο τέλος. Ο κύριος Λόχη τώρα από τη Φιλανδία έχει το λόγο. Ευχαριστώ και η Φιλανδία θεωρεί το σύστημα αυτό, τη CCTV δηλαδή, και τους στόχους, ε, κάτι που θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε. Οι διακρατικές δραστηριότητες πρέπει να γίνουν πιο απλές για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς για τις επιχειρήσεις και για την αποφυγή του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού. Βέβαια, εδώ μιλάμε για μια ευρεία εναρμόνιση της φορολόγησης εταιριών που εγείρει ερωτήματα, ιδίως όπως υπόθηκε και προηγουμένως, το γεγονός ότι οι διασυνοριακές ε, απώλειες ε, πώς αντισταθμίζονται στο μέλλον θα πρέπει να φορολογείται ε, το κέρδος εκεί που παράγεται και δεν ξέρω κατά να έχει βρεθεί η σωστή φόρμουλα. Τι γίνεται με τα άλλα αγαθά δεν λαμβάνονται υπόψη. Πού δημιουργείται η αξία, πού παράγεται η αξία, δεν είναι σαφές. Οι ιδέες πάντως οι οποίες έχουν παρουσιάσει εδώ οι συγητές, παραδείγματος χάρη ότι και η ψηφιακή οικονομία πρέπει να συμπεριληφθεί, είναι κάτι που μπορούμε να υποστηρίξουμε. Θα τις στηρίξουμε αυτές τις ιδέες. Για την Google, τη Facebook επίσης συμφωνώ και εγώ, δεν έχουν πληρώσει τους φόρους που τους αναλογούν. Πρέπει να τα διορθώσουμε αυτά τα κακοσκήμενα. Επίσης θέλω να πω ότι όταν ο στόχος είναι να δημιουργήσουμε αυτά τα δύο συστήματα, αλλά να εντάξουμε και, και τι μεγάλε εταιρείε, φοβόμαστε πω αυτό δημιουργήσει μεγαλύτερη γραφειοκρατία. Επειδή ακριβώ υπάρχουν δύο συστήματα διαφορετικά. Οι στόχοι δηλαδή είναι θετικοί, και αξιέπαινη. Παραδοσιακό όμω τα στήματα αυτά είναι εθνική κυριαρχία, εθνική αρμοδιότητα και τα φορικά και, το, και τα περί ανταγωνισμού. Ευχαριστώ πολύ. Μπράιν Χέις από Εσείς δεν φεύγετε από ό,τι ξέρω τουλάχιστον. Ε, το παρόν δεν έχω τέτοια σχέδια, λέει ο κύριος Χέις. Το τελευταίο θέμα που τέθηκε από τους συναδέλφους των Εθνικών Κοινοβουλίων είναι βασικό. Μένει να γίνει πάρα πολύ δουλειά ακόμα και δεν θα πρέπει να βιαζόμαστε γιατί οι ανησυχίες που εκφράστηκαν είναι σαφείς. Υπάρχουν δύο βασικές αρχές. Πρώτον, κανένα κράτος μέλος δεν θα πρέπει να υποχρεωθεί να κάνει κάτι το οποίο πιστεύει ότι είναι εις βάρος του εθνικού του συμφέροντος και συμφωνώ με αυτά που είπε ο κ. Λαμασό προηγουμένως για την αρχή της ομοφωνίας η οποία θα πρέπει να εφαρμόζεται για την συγκεκριμένη πρόταση. Κανένας δεν μπορεί να υποχρεωθεί, να αναγκαστεί να κάνει κάτι τέτοιο. Δεύτερον, καμία χώρα δεν μπορεί να κάνει κάτι το οποίο πιστεύει ότι θα μειώσει τη φορολογική του βάση. Και αυτό είναι το θέμα εδώ. Πολλοί συνάδελφοι είπαν ότι δεν υπάρχει μεγάλη αξιοπιστία στις εκτιμήσεις οι οποίες έχουν γίνει για το τι συνέπειες θα είχε ε, κάτι τέτοιο για τη δική μου χώρα, την Ιρλανδία. Εμείς εισπράττουμε 7,5 δις εταιρικό φόρο. Τα μισά από αυτά προέρχονται από 10 επιχειρήσεις, 10 πληρωτές, 10 μεγάλες επιχειρήσεις που ήρθαν στην χώρα μας έχουν προσλάβει ε, δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, ε, πραγματικούς πολίτες, δεν είναι ε, γραμματοκιβώτια οι εταιρείε αυτές και το 2 τρίτα από αυτές τις εταιρείε θα επηρεαστούν αρνητικά, κάτι το οποίο θα είναι μια ζημία για την Ιρλανδική οικονομία. Συνεπώς λοιπόν είναι κάτι το οποίο φύγει τις μικρές χώρες με υψηλά βιομηχανοποιημένες κοινωνίες. Κυρία Μπερέζη σας άκουσα και θα σας ακούσω μάλλον όταν έρθει η στιγμή. Συνεπώς λοιπόν, ξέρετε ότι οι οικονομίες μας έχουν περάσει από διαδικασίες μετασχηματισμού και έχουν ανάγκη τις σημερινές τους δραστηριότητες. 7,5 δις λοιπόν εισπράττουμε. Πρέπει να προσπαθήσουμε έτσι ώστε τα κοινοβούλια των κρατών μελών που ακούστηκαν σήμερα θα πρέπει να εισακουστούν και σε αυτό εδώ το κοινοβούλιο. Οι απόψει των κοινοβουλίων των κρατών μελών δεν μπορεί να αγνοηθεί από τις πλειοψηφίες που δημιουργούνται σε αυτό εδώ το κοινοβούλιο. Ακόμα και οι μειονοτικέ, αν θέλετε, μειοψήφικε συγγνώμη φωνέ θα πρέπει να ακούγονται σε αυτό εδώ το κοινοβούλιο. Γιατί υπάρχει η αντίληψη ότι ορισμένες μεγάλες χώρες κυνηγούν κατά κάποιο τρόπο τις μικρές και τέλος, ε, για τον φορό για τις ψηφιακές ε, συναλλαγές. Δεν βασίζεται στην αξιολόγηση ε, της, του κέρδους, αλλά του κύκλου εργασιών. Νομίζω ότι αν κάτι τέτοιο πράγματι ισχύει, είναι κάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει τις μεγάλες επιχειρήσεις που μπορούν να απορροφήσουν τις ζημίες και όχι τόσο τις μικρές επιχειρήσεις. Συνεπώς λοιπόν είναι κάτι, ένας φόρος που θα επιβληθεί σε ένα τομέα της οικονομίας που κυριαρχείται από επιχειρήσεις που ανήκουν στις Ηνωμένε Πολιτείες της Αμερικής. Και αυτό θα θεωρηθεί σαν μια αντι, θα έλεγα, ανταγωνιστική λήψη μέτρων. Ευχαριστώ. Πρέπει να ακουστούμε. Ευχαριστώ πολύ. ένα από Δανία, αν δεν κάνω λάθος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Χωρίς μικρόφωνο η ομιλήτρια. Er, øh, η δική μου χώρα νομίζω ότι μπορεί να συγκριθεί με τις χώρες στις οποίες αναφέρθηκαν οι προηγούμενοι συνάδελφοι. Μικρές χώρες ε, στραμμένες στην εξαγωγή. Νομίζω ότι με τον κανονισμό αυτό θα χάσουμε αρκετά χρήματα. Παρ' όλα αυτά, εν πωλής στηρίζουμε κάποιες από τις προτάσεις αυτές. Είναι ένας κανονισμός ο οποίος μπορεί να αντισταθμιστεί στην αρχή εφαρμογής του και το υποστηρίζουμε γιατί θα πρέπει να σταματήσουμε το παιχνίδι το οποίο ακολουθούν ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες για λόγους που αυτές ξέρουν Θυμίζω ότι μια επιστολή της κυβέρνησης της Δανίας ε, ε, παρουσιάζει τις θέσεις μας που στηρίζει η πλειοψηφία των κομμάτων σχετικά με τον σεβασμό της αρχής της επικουρικότητας. Αυτό είναι το βασικό. Αυτό θα πρέπει να επιδιώξουμε. Η αρχή της ε, επικουρικότητας εδώ δεν είναι κάτι το απλά τυπικό. Το θέμα είναι να δούμε αν έχουμε μια κάποια κυριαρχία σε εισαγωγικά επί των κεφαλαίων των πολυεθνικών επιχειρήσεων, κάτι το οποίο δυστυχώς δεν συμβαίνει. Αυτού του είδους τα κεφάλαια δεν κυκλοφορούν με διαφανείς τρόπους. Συνεπώς λοιπόν δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε αυτό και θα πρέπει να καταλήξουμε σε ένα μοντέλο χρήσιμο για όλους. Αυτό το οποίο είναι βέβαιο σήμερα είναι ότι υπάρχει φορολογική απάτη. Υπάρχει μη πληρωμή φορολογικών εσόδων. Εμείς δεν έχουμε εξετάσει σε βάθος την πρόταση η οποία γίνεται, θεωρούμε όμως ότι βελτιώνει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι επακριβέστερη. Το θέμα δεν είναι όμως μόνο η φοροδιαφυγή, υπάρχουν και άλλα θέματα, υπάρχουν και άλλες φορολογικές απάτες που θα πρέπει να μας απασχολήσουν. Θα πρέπει επίσης να στηρίξουμε και το λεγόμενο τέταρτο σετ κριτηρίων. Η Δανία έχει ένα, μια βάση φορολογική ευρυτάτη. Αυτό σημαίνει ότι οι προτάσεις αυτές αν γίνουν δεκτές θα την μικρύνουν, θα την πραγματικά συρρυκνώσουν. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει λοιπόν να το συζητήσουμε. Δεν ξέρουμε τις τελικές προτάσεις. Δεν ξέρουμε το τελικό αποτέλεσμα της διαδικασίας την οποία συζητάμε και εξετάζουμε σήμερα ε, σχετικά με τις μειώσεις που γίνονται στον τομέα της έρευνας ε, των, ε, της και ανάπτυξης. Συνεπώς διαρωτώμεσα εάν πράγματι οι προτάσεις που γίνονται είναι οι καλύτερες δυνατές. Εν πολλής θα συμφωνήσω και με αρκετούς Ιρλανδούς συναδέλφους, ο δρόμος που μένει να διανυθεί είναι μακρύς, αλλά σχετικά με αυτά τα οποία πιστεύει το κόμμα μου, ε, νομίζω ότι οι προτάσεις αυτές μπορούν εν πολλής να γίνουν σεβαστές. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπαλαούρας έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαστε σύμφωνοι για θέσπιση κοινών κανόνων προσδιορισμού κοινή βάση φορολογία εταιρεών που ανήκουν σε πολυεθνικούς ομίλους. Πρέπει να σημειώσω ότι ιδιαίτερα στην Ελλάδα υπάρχει πολλή φοροδιαφυγή και έχουν κυκλοφορήσει λίστες όπως η περίφημη λίστα Φαλτσιανή που στην Ελλάδα τη λέμε λίστα Λαγκάρντ όπως και λίστα Μπόγιανος από τον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών της Βεσφαλίας. Ε, πρέπει λοιπόν να υπάρξει πολλή δουλειά ακόμα αλλά και πολλή αποφασιστικότητα. Ακούω τους συναδέρφους που μίλησαν προηγουμένως και μου κάνει εντύπωση το εξής ότι ενώ οι πολυεθνικές πληρώνουν το 1 τρίτο μόνο από, αυτά που πληρώνει ένα μικρό βιβλιοπωλείο, ένα μπακάλικο, ένα ε, ε, ε, μικρό μεταποιητικό εργοστάσιο, μια μικρομεσαία ε, επιχείρηση αγροτικών προϊόντων. Δεύτερον, θέλω να πω ότι ε, στα επιμέρους ζητήματα θα πρέπει να μην τροποποιηθεί η μείωση του ορίου των 750 εκατομμυρίων στο ποσό όπως υπάρχει πρόταση στα 40 εκατομμύρια για την κοινή βάση φορολογίας των εταιριών. Τρίτον, συμφωνούμε με την, με την προτινόμενη μείωση της, πρόθετης... της πρόσθετης έκπτωσης των δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη στο 33% ώστε να στηριχτεί η καινοτομία και η οικονομία χωρίς υπέρμετρη ε, μείωση των φορολογικών εσόδων. Τέλος, υπάρχει θέσπιση της διάταξης ε, για την έκπτωση φόρου για την ανάπτυξη και επενδύσεις, η οποία θα επιφέρει θετικά αποτελέσματα, δεδομένου ότι θα συμβάλλει στη μείωση του χρέους των εταιριών και κατά συνέπεια στη μείωση των κινδύνων που απο, απο, ε, από το υποβολικό χρέος. Θα ήθελα να σημειώσω τέλος ότι για την ψηφιακή οικονομία δεν αφορά μόνο τις ε, εταιρείε οι οποίες θα εφαρμόσουν μόνο αυτό το, τον κανόνα, αλλά είναι πολύ ευρύτερο το πλαίσιο να, πω μόνο κάτι το οποίο έχει γραφτεί επανειλημμένα και έχει εντυπωσιακό ε, αποτύπωμα. Ποιο είναι ότι η Google και η Apple απέφυγαν να πληρώσουν 5 δισεκατομμύρια ευρώ στην τελευταία τριετία μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατανοείτε λοιπόν ότι εδώ υπάρχει μια τεράστια τρύπα φορολογικών εσόδων που πρέπει αποφασιστικά αν θέλει και σε αυτό το πεδίο να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι δυνάμεις οι οποίες παίζουν το μεγαλύτερο ρόλο σε αυτήν την ε, ενότητα. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much and uh, thank you for excellent... Ευχαριστώ και εξαιρετικό ήσασταν και στη διαχείριση του χρόνου αγόρευση. Σα ευχαριστώ και γι' αυτό. Τώρα περνάμε στην Αυστρία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην κυρία Ρέγνερ που είναι και η σκιώδηση στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Επιτροπή Γιούρι, όπως τη λέμε εδώ, που ήδη ψήφισε την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω και να στραφώ στον Τσέχο συνάδελφο. Την δεκαετία του 1935 και είναι 29% σήμερα. το ποσοστό φορολογίας. Ε, βέβαια θα ήταν καλό να βάλετε ακουστικά σας για να με ακούσετε γιατί θα μιλήσω ε, τώρα στα γερμανικά. Εγώ... Κοιτάξτε, θα πρέπει... Εμείς, ε, να σας πω ότι εμείς ψηφίσαμε ήδη στην Βουλή μας, οπότε θα ήθελα να αναφέρω κάποια στοιχεία με τα οποία συμφώνησαν ε, οι βουλευτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρώτα απ' όλα ψηφίσαμε και η πλειοψηφία συμφώνησε ότι πρόκειται περί ενός πακέτου, δηλαδή ότι πάει μαζί ε, με την κοινή βάση και η ενοποίηση. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ο ορισμός ε, του τι εννοούμε ψηφιακή έδρα. Ξέρουμε πως οι επιχειρήσεις σήμερα έχουν την δυνατότητα διασυνοριακής λειτουργίας ε, μέσω των ψηφιακών μέσων και έχουμε τις συστάσεις BEPS 1 ε, του ΩΣΑ και εκεί πέρα βρήκαμε τους σχετικούς ε, ορισμούς και θεωρούμε ότι αυτό θα πρέπει να υπάρχει στην τελική ρυθμισή. Κάτι άλλο το οποίο θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και το εγκρίναμε κατά βλοψηφία στο Κοινοβούλιο είναι το όριο των 40 εκατομμυρίων να παραμείνουμε δηλαδή στον ορισμό της οδηγίας, δηλαδή να μιλάμε για επιχειρήσεις που είναι πραγματικά μεγάλες και ξεπερνούν τα 40 εκατομμύρια και τέλος θα ήθελα να τονίσω τις εξαιρέσεις για έρευνα και ανάπτυξη. Εδώ πέρα θα πρέπει να υπάρχουν δημόσιες επιδοτήσεις και όχι φοροαπαλλαγές όπως προτείνει η Κομισιόν. Συνολικά λοιπόν πηγαίνει η πρόταση προς μια προοδευτική θέση και αυτό ακριβώς ε, αναζητούμε και πρέπει να ληφθεί υπόψη στην συζήτηση εθνική και ευρωπαϊκή διάσταση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κατόπιν από την Ιταλία, ο κύριος Γκουερέρη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω πρώτα απ' όλα ότι είμαστε υπέρ ε, και στηρίζουμε το περιεχόμενο της πρότασης. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι χρησιμοποιούμε απερχιωμένα εργαλεία και μονομερή μέτρα για να αντιδράσουμε στις προκλήσεις της ε, ψηφιοποιημένης και παγκοσμιοποιημένης ε, οικονομίας. Βλέπετε ότι τα κέρδη μπορούν να καταγραφούν σε διάφορα μέρη με έναν συνδυασμό επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και βεβαίως έχουμε κέρδη που δεν ε, συνδέονται με κάτι το απτό, όπως παραδείγματος χάρη αυτά τα οποία προκύπτουν από την πνευματική ιδιοκτησία. Πρέπει λοιπόν να προσαρμόσουμε την φορολογία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να είναι δίκαιη και λιγότερο κατακαιρματισμένη στην ενιαία αγορά. Θα πρέπει λοιπόν να στηρίξουμε τις ε, προτάσεις και τις δύο. Η Ευρωπαϊκή Συνεργασία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη ήταν ανεπαρκής και συναντά την κριτική και την αδιαλαξία ορισμένων κρατών μελών. Δεν πείθουν όμως τα αντεπιχειρήματα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να επιμείνουμε και να ξεκαθαρίσουμε ότι κοινή φορολογική βάση δεν σημαίνει πως η χώρα θα πρέπει να φέρει έναν ελάχιστο εθνικό φορολογικό συντελεστή, ούτε ότι δεν θα μπορούν να ανταγωνίζονται με χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές. Αυτό το οποίο ισχύει είναι ότι μια κοινή πανευρωπαϊκή βάση θα κλείσει πολλά παράθυρα για τις πολυεθνικές για να χειραγωγούν την φορολογική τους θέση. Επιπλέον, μια κοινή ενοποιημένη βάση φορολογικής επιχειρήσεων, αυτό φορολογητέο κέρδος θα μπορεί να μοιραστεί μεταξύ των χωρών όπου λειτουργεί μια εταιρεία ανάλογα με τον τζίρο στην εν λόγω χώρα και τον φορολογικό συντελεστή. Και έτσι βεβαίως και οι εταιρείε θα το στηρίξουν γιατί μειώνεται το κόστος συμμόρφωσης και από την άλλη πρέπει να πούμε ξεκάθαρα πως η κοινή φορολογική βάση θα αυξα... θα αυξήσει, δεν θα μειώσει τον ανταγωνισμό μεταξύ των κρατών μελών. Γιατί αν υπήρχε πραγματικά μια εναρμονισμένη κοινή φορολογική βάση, θα υπήρχε πίεση στους φορολογικούς συντελεστές προς τα κάτω. Αυτό το επιβεβαιώνουν και τα στοιχεία. Και τούτου λεχθέντος νομίζω ότι είναι σημαντικό και στηρίζω την ιδέα μιας ε, σοβαρής αξιολόγησης αντικτύπου που πρέπει να εφαρμοστεί και να ενισχυθεί στο μέλλον. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Από την Μάλτα ο κύριος Μπούσουτιλ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να συμφωνήσω με τους συναδέλφους από την Ιρλανδία και την Κύπρο που εξέφρασαν ε, την αντίθεσή τους με τις προτάσεις αυτές. Όπως και εκείνη. θεωρώ ότι αυτές οι προτάσεις πρώτα απ' όλα παραβιάζουν την αρχή της επικουρικότητας. Αυτό είναι σαφώς ένας ε, τομέας που ανήκει στη φορολογία. Η φορολογία είναι εθνική αρμοδιότητα και το να περάσουμε σε αυτόν τον τομέα παραβιάζει την αρχή της επικουρικότητας. Αλλά κάτι πιο θεμελιώδης θεωρώ ότι οι προτάσεις αυτές ε, θα επηρεάσουν αρνητικά τις οικονομίες κάποιων χωρών. Θα υπάρχει σοβαρός αντίκτυπος στα φορολογικά έσοδα και στην απασχόληση και στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Δεν μπορούμε απλά να λέμε ότι αυτά τα πράγματα δεν θα γίνουν επειδή δεν το θέλουμε. Αυτά είναι σοβαρές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κάποια κρατημέλη και προτείνω να τα πάρουμε σοβαρά. Υπάρχει μια πρόταση να υπάρξει κάποιο ταμείο αποζημίωσης για να βοηθήσουν αυτούς οι οποίοι θα επηρεαστούν αρνητικά από αυτές τις προτάσεις. Αλλά αναρωτιέται κανείς γιατί να προξενήσουμε τη ζημία και μετά να δώσουμε αποζημίωση. Ε, ξέρετε η χώρα μου κύριε Πρόεδρε είναι υπέρ τη ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στη χώρα μου ακόμα, ο κόσμος δεν μπορεί να αντιληφθεί γιατί γίνονται αυτές οι προτάσεις και γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να μπει σε αυτό το θέμα. Υπάρχει αίσθηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κάνει αρκετά σε τομείς όπου θα έπρεπε να κάνει περισσότερα, αλλά μπλέκει σε τομείς όπου ε, δεν έχει καμία δουλειά να μπλέκει. Και προφανώς αυτό οδηγεί σε κάποια αντιευρωπαϊκό συνέστημα που όλοι ξέρουμε ότι έχει οδηγήσει σε πολύ αρνητικές συνέπειες σε άλλες χώρες. Ναι, να μην πούμε τίποτα για την άνοδο λαϊκιστικών κομμάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Σαφώς ε, είναι αντίθετα πολλά κράτη-μέλη και πρέπει αυτό να το λάβουμε σοβαρά υπόψη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και περνάμε ξανά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο κ. Κάρφη από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που είπαν οι προλαλήσαντε. Απλά θα τα βάλω στο πολιτικό πλαίσιο τα πράγματα. Εγώ προσωπικά είμαι υπέρ η χώρα μου να συνεχίσει την βιώσιμη βιομηχανική προσέγγιση που δεν θα βασίζεται μόνο στην προσέλκυση των πολυεθνικών που σίγουρα βέβαια θα συνεχίσουν να παίζουν ρόλο για την μικρή μας χώρα την Ιρλανδία. Αλλά η χώρα μας δεν έχει μια κυβέρνηση που ακολουθεί αυτή τη βιώσιμη οικονομική στρατηγική. Γι' αυτό και υπάρχουν ανησυχίες από όλο το πολιτικό φάσμα για τη δυσανάλογη ε, επίδραση και την αρνητική επίδραση που θα έχει το CCTB στην οικονομία μας και στην παροχή των δημόσιων υπηρεσιών. Να σας πω για κάποιες δικές μου ανησυχίες. Η βασική είναι ότι τα κράτη-μέλη τελικά ζητούνται να μεταφέρουν εξουσίες τους στην Κομισιόν με αντάλλαγμα την υπόσχεση ότι το νέο σύστημα θα αποτρέπει τις πολυεθνικές από τη μετατόπιση κέρδους. Ουσιαστικά όμως η πρόταση λέει ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν θα επιτευχθεί αυτός ο στόχο. Σε ό,τι αφορά τώρα τη μοναδία φορολογία για την αποφυγή της μετατόπισης κερδών, αυτό θα πρέπει να γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο και πρέπει να το ξέρετε κι εσείς ότι η εφαρμογή της CCTB σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα έχει ως αποτέλεσμα μάλλον να μεταφερθούν οι απώλειες ενός κράτους και στα άλλα. Θα πρέπει μόνο ε, να έχουμε υπόψη ότι μπορεί η μετατόπιση κερδών να περιοριστεί εντό Ένωση. αν είναι η προσέγγιση ενιαία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα οξυνθεί η τάση να μεταφέρονται τα κέρδη εκτός Ευρωπαϊκή Ένωσης. Και θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τη μεταφορά των ε, δραστηριοτήτων και των κερδών ε, στις δικατορικές εκτός Ένωσης. Σε ό,τι αφορά τώρα τον ορισμό ε, της ε, Κομισιόν, για την μητρική εταιρεία, αναφέρεται ε, κάποια λύση, μερική λύση στην έκθεση των εισηγητών, αλλά με την χρησιμοποίηση των ενοποιημένων λογαριασμών μπορούν να προκύψουν πολλά ωφέλη για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Υπάρχει επίσης μια μελέτη η οποία δείχνει ότι οι βάσεις φορολογίας μειώνονται. Και δεν νομίζω να αλλάξουν τα πράγματα αν υπάρχει αυτή η αλλαγή προσέγγισης. Επίσης ανησυχώ και για το τι θα, κάνει, τι θα γίνει με την οδηγία για κατά της φόρο αποφυγής, όπως είπαν και άλλοι προλαλήσαντες. Αν μου επιτρέπετε τέλος, από το πολιτικό φάσμα συνολικά νομίζω ότι πρέπει να στηρίξουμε την μοναδία πρόταση για τα μέτρα φορολόγησης. Αυτό νομίζω ζητούν οι φορολογούμενοι και εμείς πρέπει να το στηρίξουμε. Thank you. Uh, next από την Πορτογαλία ο επόμενος ομιλητής, ο κ. Περέιρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να πω ποια είναι η άποψη του Πορτογαλικού Κοινοβουλίου. Εγκρίθηκε μια έκθεση και από την Επιτροπή Προπολογισμού, εγώ είμαι αντιπρόεδρος της, με παρόδο, και από την Επιτροπή για τα Ευρωπαϊκά Ζητήματα, τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις. Και η έκθεση αυτή είναι εν γέννη υπέρ της κοινή γενοποιημένη βάση φορολόγηση εταιριών. Πρώτον, γιατί θεωρούμε ότι σέβεται την αρχή της επικουρικότητας, με τον πολύ απλό λόγο, ότι ο στόχος αυτός δεν θα μπορούσε αποκεντρωμένα συγγνώμη, να επιτευχθεί. Δηλαδή αναχώρα. Καλό είναι λοιπόν να υπάρχουν οι ίδιοι κανόνες για τη βάση φορολογής επιχειρήσεων. Δεν είναι κάτι ανέφικτο. Θα πρέπει να γίνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωσης λοιπόν. Και η αρχή της αναλογικότητας γίνεται σεβαστή. Δηλαδή τα μέτρα που προτείνονται κρίνονται απαραίτητα για την επιτεύξη των στόχων και αναλογικά. Άρα κατά βάση είμαστε υπέρ. Βέβαια, Υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορούν και πρέπει να συζητηθούν, όπως είναι το κατόφλι. Τα 750 εκατομμύρια είναι πολύ ψηλό. Θα πρέπει να είναι χαμηλότερο το κατόφλι, πιστεύουμε. Επίσης, μάλλον δεν έχω και πολύ χρόνο, άρα να συνοψίσω λίγο. Αλλά επειδή Άκουσα και κάποιους προλελήσαντες ε, να εκφράσουν τις απόψεις τους. Θέλω να πω και εγώ τη δική μου άποψη. Η Ιρλανδία μίλησε. Σαν οι μικρές χώρες όλες να έχουν την ίδια άποψη. Εμείς είμαστε μικρή χώρα, αλλά έχουμε διαφορετική άποψη. Άρα δεν έχουμε να κάνουμε μικρές μεγάλες χώρες. Σίγουρα πρέπει να ακουστούν προσεκτικά όλα τα επιχειρήματα. Αλλά θα πρέπει να δούμε καταρχάς τη μεθοδολογία. να μην τα συζητούμε μέσα σε ένα πέπλο άγνοια. Δηλαδή, πρώτα πρέπει να έχουμε μια μελέτη αντικτύπου. Και αυτό θα ήταν το δεύτερο βήμα. Το πρώτο βήμα είναι να αρχίσουμε να συζητούμε. Το κατά πόσο είναι δίκαιο και θεμητό διαφορετικές χώρε να έχουν διαφορετικούς τρόπους υπολογισμού των φορολογικών εσόδων. Και αν αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την φόρο αποφυγή ή για το φορολογικό, επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό από κάποιε επιχειρήσει. Θα γίνει πρώτα η συζήτηση και ενδεχομένως καταλήξουμε σε κάποιες κοινέ αρχές. Και αν γίνει αυτό, θα πάμε στο δεύτερο βήμα, που είναι η μελέτη αντικτύπου, για να δούμε ποια χώρα και ποιο τομέα χάνει και γιατί. Και όχι μόνο πόσο χάνει, αλλά γιατί χάνει. Ιρλανδία. Απλά χρησιμοποιώ το παράδειγμα της Ιρλανδίας, είναι πιο απλό. Τι φταίνει οι κανόνες της ε, βάσης ε, φορολόγησης επιχειρήσεων ή φορολογικοί συντελεστές. Ήταν πολύ χαμηλός φορολογικός από πάρα πολλά χρόνια και γι' αυτό ωφελούνταν. Δεν είμαι και βέβαιος βέβαια, θα ήθελα να δω τη μελέτη. Γιατί θα χάσουν. Γιατί έγινε λόγος ότι θα χάσουν και ίσως και 5%. Γιατί θα χάσουν οι χώρες, πόσο θα χάσουν, αυτό είναι κάτι που πρέπει να το μελετήσουμε. Και ολοκληρώνω με το εξή. Νομίζω ότι αυτό το Ταμείο αντιστάθμισης του κ. Λαμασούρ θα είναι απαραίτητο. Γιατί φυσικά οι χώρες που θα χάσουν, και αυτό θα, θα πρέπει να φασιστεί με ομοφωνία, θα πρέπει να αντισταθμίζονται, να αποζημιώνονται με κάποιο τρόπο. Και αυτό το ταμείο θα βοηθήσει, πιστεύουμε. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, πριν δώσω τώρα το λόγο στον επόμενο μιλητή, να σας πω ότι θα είναι ο τελευταίος ε, από τα Εθνικά Κοινοβούλια και θα έχουμε και άλλους δύο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είμαστε μέσα στο χρόνο. Οπότε ακόμα και αν κανένα δύο ακόμη θέλετε το λόγο μπορούμε να σας συμπεριλάβουμε στον κατάλογο. Αλλά μένουν τρεις. Τελευταίες από τα Εθνικά Κοινοβούλια, ο κύριος Κράινερ από την Αυστρία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε από σε λεπτομέρειες για... Νομίζω ότι όλα αυτά έχουν υπογραμμιστεί που θα ήθελα να πω και από άλλους συναδέλφους. Θα ήθελα εγώ να ζητήσω ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα κοινό ελάχιστο, μια κοινή ελάχιστη επιβολή, ε, όπως επίσης και η λεγόμενη φορολογική οδή, η διάδρομη αν θέλετε, Νομίζω ότι δεν μπορούμε να γνωρίσουμε την πραγματικότητα η οποία λέει ότι η φορολογία αυξάνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια. Και αυτό σημαίνει ότι αυτοί οι οποίοι βολεύονται με την κατάσταση αυτή είναι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις και πάρα πολύ πλούσιοι άνθρωποι. Και τα σχολεία δεν είναι τόσο καλά, τα νοσοκομεία δεν είναι τόσο καλά γιατί η κοινωνία και το κράτος δεν είναι σε θέση να κάνει αυτά τα οποία πρέπει συνεπώς λοιπόν αυτοί οι οποίοι έχουν, αυτοί πρέπει να πληρώνουν και δεν θα πρέπει να φορολογούνται συστηματικά και αποτελεσματικά μόνον οι α, μεσαίες τάξεις. Λοιπόν, ναι CCTV, αλλά με μειωμένα ποσοστά επιβολής φόρου από τη μία και τους λεγόμενους φορολογικούς διαδρόμους από την άλλη. Και έτσι οι χώρες όπως η Αυστρία ή και άλλες χώρες οι οποίες δεν χρειάζεται να προλάβουν κάποιο άλλο επίπεδο θα μπορέσουν να συνεχίσουν να λειτουργούν ικανοποιητικά. Τώρα για την αρχή της επικορικότητας. Έχουμε το κοινοτικό επίπεδο, το εθνικό επίπεδο και το ευρωπαϊκό επίπεδο. Συνεπώς, ανάλογα με την πολιτική που θέλει να εφαρμόσει κανείς, το θέμα είναι ποιος είναι υπεύθυνο και σε ποιο επίπεδο είναι πιο αποτελεσματική η ευθύνη η οποία αυτή πρέπει να ασκηθεί. Συνεπώς λοιπόν χώρες οι οποίες δραστηριοποιούνται σε 2, 3 ή 20 ευρωπαϊκές χώρες είναι σαφές ότι ο τρόπος φορολογίας τους είναι κάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία και είναι σαφές ότι θα πρέπει να εφαρμόζεται η φορολογία σε ευρωπαϊκό επίπεδο γιατί ακριβώς λειτουργούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ακόμα και σε επίπεδο αρχής επικουρικότητας μπορούμε να δεχθούμε ότι οι ευρωπαϊκές εισαγωγικά επιχειρήσεις πρέπει να φορολογούνται ευρωπαϊκά. <coughs> έχουμε και ένα εκπρόσωπο του Σοσιαλιστικού Κόμματος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Has Έχουν τροχιαστεί οι προσπάθειες ε, καταπολέμησης της ε, φόρο και επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού ανταυτού. Ο πραγματικός στόχος έχει γίνει ο περιορισμός του φορολογικού ανταγωνισμού για να πάμε προς μία εναρμόνιση. Μα εδώ πέρα βάζουμε το κάρο μπροστά από το άλογο. Οπωσδήποτε βεβαίω, ο φορολογικό ανταγωνισμό χρειάζεται στι μικρέ χώρε στην Ιρλανδία και τι ε, άλλε για να μπορέσουν να αντισταθμίσουν τα μειονεκτήματά του όπω η απόσταση από τι μεγάλε αγορέ επιπλέον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τι περιορίζει με του όρου του Συμφώνου σταθερότητα και οι χώρε οι οποίε έχουν μειώσει του συντελεστέ ε, υπερβολικά πρέπει να βρουν άλλου ε, πόρου. Το να πηγαίνουμε προς την ε, φορολογική εναρμόνιση. Πρώτα, μια κοινή βάση φορολογίας ε, εταιρείων δεν στέκει και για πολιτικούς και για οικονομικούς λόγους. Ακόμα και η ΕΠΑ, ένα ομοσπονδιακό κράτος, δεν έχει κάτι τέτοιο. Και μάλιστα, ήδη, σήμερα με τους περιορισμούς του Δημοσιονομικού Συμφώνου, τα κράτη-μέλη έχουν περισσότερους ε, περιορισμούς προπολογισμού τους από ότι οι πολιτείες των ΕΠΑ. Θα πρέπει λοιπόν τα κράτη-μέλη ασκώντας την κυριαρχία τους να κάνουν περισσότερα για να καταπολεμήσουν την κατάχρηση των ε, φορολογικών συστημάτων και μάλιστα καλό θα ήταν να υπάρξει μια ανταλλαγή πληροφοριών ε, ειδικά με τις είπα όπως ε, κάνουν εκεί με η νομοθεσία η οποία λέγεται ΦΑΤΚΑ. Οπότε δεν αντιλαμβάνομαι γιατί οι εθνικές φορολογικές διοικήσεις δεν πάνε πάρα πέρα και δεν δημοσιεύουν πλήρως ε, καταλόγους ατόμων και επιχειρήσεων ε, με τους φόρους που πλήρωσαν. Έτσι θα υπάρχει ένας δείκτης ο οποίος θα μας δείχνει το τι συνέβη και σε εθνικές αγορές και σε διασυνοριακό επίπεδο και έτσι μπορούμε να τα διασταυρώσουμε αυτά μέσω του ΦΥΠΙΑ. Εάν είναι αναγκαίο ας βελτιώσουμε το καθεστώς του ΦΥΠΙΑ. Και βεβαίως ο μέσος όρος των συντελεστών ανακλάδο ή αποτελεί ένα άλλο εργαλείο. Και πάντα βεβαίως μπορεί το κράτος να επιβάλλει φόρο κύκλου συναλλαγών ε, για να φορολογήσει τα κέρδη. Να πω λοιπόν το εξή για να καταπολεμήσουμε την κατάξυση των φορολογικών συστημάτων. Δεν έχουμε εξαντλήσει τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Το να ίσκουμε τώρα νέα μέσα είναι αντιπαραγωγικό και βεβαίως κατά των συμφερόντων κάποιων κρατών μελών. Ο στόχος στο ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να είναι η διαφάνεια και στο ευρωπαϊκό επίπεδο και στο επίπεδο του ΩΣΑ. Now, uh, Ευχαριστώ, Ακούμε πολλούς συναδέλφους, πολλοί από αυτούς λένε τα ίδια πράγματα, κάποιοι άλλοι διαφοροποιούνται. Μου κάνει εντύπωση το περιεχόμενο των συζητήσεων που ακούσαμε εδώ. Είναι σαν να, να είχαμε καταθέσει μια πρόταση βιαστική, μια πρόταση ε, με το ζόρι να την είχαμε καταθέσει, ενώ θα έπρεπε να δουλέψουμε πάνω σε αυτή ακόμα περισσότερο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Από την άλλη, υπό την πίεση των εκλογών μας και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το θέμα της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και της φορολογικής απάτης έχει προχωρήσει ακόμα και στο Συμβούλιο και έχουν εξεμπλοκάρει ορισμένα ντοσιά. Η ιδέα λοιπόν του να περάσουμε σε αυτό το νέο CCTB είναι κάτι που ανταποκρίνεται σε αυτήν την περιγραφή την οποία έκανα προηγουμένως. Δεν θέλω να μιλήσω για την πτωχοποίηση των κρατών μελών, αλλά ξέρετε ότι οι χώρες σήμερα δυσκολεύονται να χρηματοδοτούν τις δημόσιες υπηρεσίες τους, έχουν προβλήματα να καταπολεμούν α, τις ανάγκες που έχουν, διότι οι επιχειρήσεις δημιουργούν νέους τρόπους παραγωγής. Μου κάνει επίσης εντύπωση Ε, το ότι δεν λαμβάνετε ίσως κάποια από εσάς υπόψη είναι ότι δεν είναι κάτι το καινούριο αυτή η πρόταση την οποία κάνουμε. Είναι η δεύτερη ε, στη σειρά. Θυμάστε την εργασία της κυρίας Πριμαρόλο. Θυμάστε ότι πριν από τη φορολογία των επιχειρήσεων υπήρχε μια κάποια μορφή ε, στρέβλωσης του ανταγωνισμού ανάμεσα στα κράτη-μέλη και εδώ να θυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάρα πολύ σωστά περιγράφει τις συνέπειες αυτής της κατάστασης. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν μετά από τη συζήτηση που άκουσα πού θέλετε να πάμε. Βλέπω ότι όταν συναντώμεθα και όταν ξαναβρεθούμε μάλλον για την διάσκεψη για το άρθρο 13 στο Ταλίν σε λίγο καιρό, ένα από τα θέματα το οποίο επέλεξε η Προεδρία αφορά μια πιο αποτελεσματική συλλογή των φόρων, εισπραξή των φόρων. Εφόσον λοιπόν αυτό είναι ο στόχος, θα πρέπει ο καθένας στο χώρα του να κινητοποιηθεί έτσι ώστε να καταλήξουμε σε καλύτερα αποτελέσματα επί τη βάση της χρήσιμης πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εδώ να σας εκφράσω την ανησυχία μου βλέπω το τι συμβαίνει στη χώρα μου και όχι μόνο στη χώρα μου. Είμαι ευρωβουλευτής αλλά βλέπω βέβαια το τι συμβαίνει στη χώρα μου και διαπιστώνω ότι υπάρχει μια πρόταση για ένα νέο φόρο για τις επιχειρήσεις σε μια βάση γαλλογερμανική. Αυτή τη στιγμή κάτι τέτοιο δημιουργηθεί στο εσωτερικό της ε, αγοράς, στα πλαίσια της εσωτερικής αγοράς, τότε η συζήτηση θα γίνει κάτω από εντελώς διαφορετικές συνθήκες. Νομίζω λοιπόν ότι έχουμε κάθε συμφέρον να συζητήσουμε το θέμα αυτό σε κοινοτικό επίπεδο, με βάση τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σύμφωνα και με αυτά τα οποία μας είπαν οι δύο συνεισηγητές, το θέμα της ε, φορολογίας των επιχειρήσεων θα τεθεί και στα πλαίσια ε, της ψηφιακής οικονομίας. Νομίζω ότι η σωστή επικουρικότητα μπορεί να λειτουργήσει στο ευρωπαϊκό επίπεδο και η σωστή συμπληρωματικότητα σημαίνει να ανακτήσουμε κάποια περιθώρια καλύτερης φορολογίες και σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σας ευχαριστώ πολύ. Πριν δώσω το λόγο στους εισηγητές θα ήθελα και εγώ να κάνω κάποιες σύντομες παρατηρήσεις. Είναι σαφές ότι υπάρχουν αρκετές ανησυχίες. Πολλοί από εμά και πολλοί οικονομολόγοι θεωρούν ότι χρησιμοποιούν την φορολογία όχι σαν κίνητρο για τις επενδύσεις, αλλά για να πάρουν χρήματα από τους προϋπολογισμούς άλλων χωρών. Λοιπόν, κάτι τέτοιο δεν μπορεί να υποστηριχθεί σοβαρά. Το δεύτερο το οποίο πρέπει να πω ότι δεν είναι μια προσπάθεια αυτό που κάνουμε για εναρμόνιση της φορολογικής μεθόδου και να τελειώσουμε την εθνική, να ανατρέψουμε την εθνική φορολογία. Νομίζω ότι η πρόταση αυτή είναι μια εξαιρετική πρόταση, γιατί σε επίπεδο στρατηγικής δίνει την δυνατότητα στα κράτη-μέλη να μετασχηματίσουν τη φορολογία τους σε ένα πιο εύκολο, αποτελεσματικό, εισπράξιμο φορολογικό σύστημα. <clears throat> Και ταυτόχρονα το κοινό θα προστατεύεται από την αύξηση της φορολογίας στην περίπτωση κατά την οποία οι χώρες έχουν ε, αδυναμία να εισπράξουν τους φόρους αυτούς και ξέρουμε επίσης ότι και η αναστάτωση που επικρατεί μερικές φορές σε επίπεδο ίσπραξης φορολογικών εσόδων φύγει τον ανταγωνισμό. Το θέμα επίσης δεν είναι ε, ε, κάτι ανάμεσα στα μικρά και στα μεγάλα κράτη. Το θέμα είναι να δούμε ποιοι χάνουν σύμφωνα με την κατάσταση που υπάρχει σήμερα. Ακούστηκε ότι θα πρέπει να ακουστούν όλες οι απόψεις και να συζητηθούν όλες οι απόψεις. Και από τις μεγάλες και από τις μεσαίες και από τις μικρές χώρες. Και από αυτές που θεωρούν ότι θα ωφεληθούν και από αυτές οι οποίες θεωρούν ότι δεν θα ωφεληθούν. Γι' αυτό λοιπόν έχω την εντύπωση ότι πρέπει να μας βοηθήσετε να κατανοήσουμε όλοι την λογική των άλλων έτσι ώστε να αποκαταστήσουμε τις γέφυρες μεταξύ μας. Εμείς θα θέλαμε να έχουμε μια καλή πρόταση, καλή για το μέλλον της Ευρώπης. Θα δώσω το λόγο όμως στους δύο εισηγητές, πέντε λεπτά ο καθένας. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους για τις ε, συνεισφορές τους, για τις παρεμβάσεις τους. Ήταν πολύ καλό που έγινε αυτή η συζήτηση. Ιδίω ήταν σημαντικό να ακούσουμε την άποψη των ε, Εθνικών Κοινοβουλίων, γιατί η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία δεν πρέπει να αποφασίζεται κάπου αλλού, αλλά και στα Εθνικά Κοινοβούλια. Και πρέπει να πω ότι προσβλέπω και στην επίθεση στην Ιρλανδία. Το θέμα δεν είναι σίγουρα μικρές μεγάλες χώρες, μπορεί να είναι μεταξύ νησιωτικών και υπηρετικών χωρών. Γιατί περισσότερε ήταν από αντιδράσεις ήταν από νησιά. Κύπρο, Μάλτα, Ιρλανδία, δεν ξέρω. Εντάξει, μπορεί να μην τα περιγράφω εντελώ πιστά τα πράγματα, αλλά η Ολλανδία, χώρα από την οποία εγώ κατάγομαι, έχει και αυτή τις ανησυχίε τη, αλλά αλλάζει και εκεί η συζήτηση, οφείλω να σας πω. Ο λόγος είναι ότι η Ολλανδία είναι σε μια μοναδική θέση, κατά κάποιο τρόπο. περί τα φορολογικά. Είμαστε μια μικρομεσαία χώρα. Αλλά είμαστε μεγάλοι σε ό,τι αφορά τη φοροαποφυγή. Νομίζω ανταγωνιζόμαστε την Ιρλανδία επαξίως. Και αυτό δημιουργεί περίεργα πράγματα. Αν δείτε τις ε, άμεσες ξένες επενδύσεις, το Λουξεμβούργο και η Ολλανδία από κοινού έχουν πολύ περισσότερες άμεσες ξένες επενδύσεις σε σχέση με την, την Αμερική της ΗΠΑ. ή από τη Γερμανία και την ε, Γαλλία, η Ιρλανδία. Τι λέει αυτό. Λέει ότι υπάρχει φορολογικός σχεδιασμός εδώ. Είναι στατιστικά. Ε, είναι τα χαρτιά που μεταφέρονται από εδώ και από εκεί. Δεν είναι πραγματικές επενδύσεις. Εγώ κατάλαβα και άκουσα πολύ προσεκτικά ότι θέλετε δημιουργία θέσεων εργασία με πραγματικές επενδύσεις. Αυτό σας ενδιαφέρει. Πραγματική δραστηριότητα, όχι στα χαρτιά. Και ακριβώς αυτή είναι η διάκριση που κάνει η πρόταση για την κοινή βάση φορολόγηση επιχειρήσεων. Άρα να σταματήσουμε αυτά τα εικονικά ε, και να, έχουμε, να προσφέρουμε πραγματικές δυνατότητες. Να εστιάσουμε με τις πολιτικές μας την πρόταση να επενδύσουμε στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Νομίζω ότι δίνει πλήστες ευκαιρίες αυτό το μέσο που προτείνουμε. Παρότι σίγουρα μπορεί να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο. Πάντως προωθεί και την ισότιμη μεταχείριση και υπάρχει και αυτή η μείωση φόρου για, φόρου για την έρευνα και την ανάπτυξη. Όσα έχει το ρόλο του να διαδραματίσει, αλλά όλο και λιγότερο θα έλεγα γιατί νομίζω ότι έφτασε στα ωριά του. Το πρώτο, σκεφτείτε το, το πρώτο σημείο του σχεδίου δράσης στον ΩΣΑ ήταν ψηφιοποίηση και έλεγε φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας. Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Πού ε, οδήγησε αυτό, πουθενά. Πέντε χρόνια ανεβλήθη και δημιουργήθηκε αυτή η task force. Γιατί, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι δεν συμφωνούν. Φυσικά, οι αμερικανικές εταιρείε, όπως είναι η Apple, το Facebook, η Google, δεν θέλουν να φορολογηθούν Άρα δεν μπορεί να γίνει κάτι εντό όσα. Άρα χρειάζεται ευρωπαϊκό ρόλο. Θα πρέπει εμεί να πάρουμε τα εννέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να περάσουμε λοιπόν σε αυτή την φορολογία όπως την προτείνουμε που πάλι θα επιτρέπει το φορολογικό ανταγωνισμό αλλά θα είναι τελείως διαφορετικός. So that's, um, let me... Uh, Δύο πράγματα, αν με επιτρέπετε, να υπογραμμίσω ακόμη. Σε ό,τι αφορά τη λογιστική, γιατί γίνεται συζήτηση. Η συζήτηση δεν αλλάζει την κατάσταση σε ό,τι αφορά τη λογιστική. Το δέχομαι όμως το σημείο. Ότι τα λογιστικά πρότυπα ίσως να είναι το επόμενο εντό εφών παιχνίδι. Δηλαδή να περνάει ο ανταγωνισμό πλέον μέσα από τα λογιστικά πρότυπα και αυτό είναι ένα θέμα που επίση πρέπει να μα απασχολήσει. Η Εύλεν Ρέγκνερ μίλησε για το κατόφλι και χαίρομαι γι' αυτό γιατί τώρα αφορά μια πολύ μικρή ομάδα, υπομάδα θα έλεγα επιχείρησεων και θα έπρεπε να καλύπτει πολύ περισσότερες. Άρα βαθμιδών θα έπρεπε να θετήσουμε μια διαφορετική προσέγγιση για να περιλάβουμε μεγαλύτερο αριθμό άρα μειώνοντα αυτό το κατόφλι. Επόμενο, σε ό,τι αφορά τη φορολογική βάση, ο Αλέλα Μασούρ, πολύ σημαντική συνεισφορά Συμφωνώ με αυτούς που είπαν ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η αξιολόγηση. Ο λόγος είναι ότι είναι πολύ δύσκολο οι Βρυξέλλες να καταλάβουν τι συμβαίνει επιτόπου στα κράτη-μέλη. Άρα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει πολύ στενή συνεργασία με τις διάφορες φορολογικές διοικήσεις για να υπάρξει αυτή η καλή αξιολόγηση που δεν έχει ακόμη σε ένα επαρκέ σημείο. Και θέλουμε να έχουμε ακριβή νούμερα, ακριβή αριθμητικά στοιχεία για τη φορολογική βάση, για, τον, για το πώ θα επηρεάσει η φορολογική βάση για τι διάφορε χώρε. Πρέπει να γίνει δουλειά πάνω σε αυτό. Τα εξετάζουμε όλα. Χρειάζεται δουλειά, πράγματι το δέχομαι, αλλά γι' αυτό απαιτείται στενή συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκή Επιτροπή και των φορολογικών διοικήσεων. Δεν μπορώ, όπω καταλαβαίνετε κύριε Πρόεδρε, να τα κάλυψω όλα. Πάντω τα σημείωσα και όποιο θέλει να έρθει σε επαφή μαζί με τα χαρά ε, να έχουμε μια πιο εντελεχή συζήτηση για πιο μεμονωμένα ζητήματα. Προς το παρόν ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση. Πρώτα σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την προσφορά που πιστεύω ότι θα την αποδεχθούν κάποιοι και τώρα το λόγο έχει ο Αλέν Λαμασούρ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους πήραν το λόγο. Σημειώσαμε αυτά τα οποία είπατε και θα ανταλάβουμε υπόψη μας. Όπως είπαν πάρα πολύ και το θύμισε και ο Πολ αυτό το οποίο μας λείπει σήμερα είναι μελέτες επιπτώσεων για να γνωρίζουμε εμείς ανά τύπο επιχείρησης και αναχώρα ποιες θα είναι οι συνέπειες της προτινόμενης μεταρρύθμισης. Προς στιγμή μιλάμε με τις μελέτες που είχαν γίνει το 2011 και από τότε έχουν πολλά αλλάξει στην οικονομία. Πολλοί από εσά αναφέρθηκαν στην αρχή της επικουρικότητας. Τι σημαίνει επικουρικότητα. Σημαίνει ότι συστηματικά τα θέματα θα πρέπει ε, να αντιμετωπίζονται συστηματικά στο χαμηλότερο δυνατό διοικητικό επίπεδο. Μήπως να μιλήσουμε για το πιο κατάλληλο επίπεδο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια σωστή διαπραγμάτευση με τις μεγάλες πολυεθνικές. Μια χώρα μπορεί να διαπραγματευτεί ισότιμα με μια μεγάλη επιχείρηση της οποίας ο κύκλος εργασιών είναι δύο φορές, τρεις φορές ή δέκα φορές μεγαλύτερο από το εσωτερικό ακαθάριστο της χώρας. Όχι βέβαια. Αν ένα θέμα λοιπόν πρέπει να αντιμετωπιστεί από κοινού σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι η φορολόγηση αυτών των γιγαντιαίων οικονομικών οντοτήτων. Άκουσα με πάρα πολύ προσοχή και αυτά τα οποία είπαν οι Ιρλανδοί συνάδελφοι, ο κύριος Οντόνελ, φυσικά εφόσον μας καλέσετε, ευχαρίστως θα είμαστε εκεί που χρειάζεται στην Ιρλανδία δηλαδή για να καταλάβουμε. Λέει ότι το σύστημα είναι διαφανές και το 12,5% είναι επίσης διαφανές. Μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Όταν η Επιτροπή λέει στην Ιρλανδία ότι θα έπρεπε να εφαρμόσετε το 12,5% στην Apple, η Ιρλανδία προσφεύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και σας παραπέμπω εδώ στην μαρτυρία του κυρίου Τιν Κούκ εδώ και δυο 3 χρόνια στην Αμερικανική Γερουσία Είχε πει τότε ο κύριος Κούκ ότι η Apple ήταν ε, ένας φορολογούμενος πρότυπο στις Ηνωμένε Πολιτείε γιατί πληρώνει για τα κέρδη που παράγει στις Ηνωμένε Πολιτείε και είπε ότι για τα κέρδη στον υπόλοιπο κόσμο που ήταν τότε το 70% έχουμε μια συμφωνία με την Ιρλανδική κυβέρνηση που μας επιτρέπει ουσιαστικά να μην πληρώνουμε. Ε, αυτό δεν θέλουμε να το βλέπουμε. Γι' αυτό ακριβώς προτείνουμε να παρακολουθούμε από κοντά το τι γίνεται στην Ιρλανδία τα τελευταία χρόνια και την κατάργηση του λεγόμενου Double Irish Tax. Για ε, αυτά τα οποία είπε ο κύριος Φίντλα θα ήθελα να σταθώ λίγο στην προσπάθεια της Γαλλίας και της Γερμανίας να ευνοήσουν τις επιχειρήσεις τους. Κοιτάξτε, οι γερμανικές επιχειρήσεις είναι τόσο ανταγωνιστικές που δεν έχουν ανάγκη από τέτοια κόλπα. Η βασική μας ανησυχία είναι να πληρώσουν οι πολυεθνικές, όχι μόνο οι αμερικανικές, αλλά κυρίως αυτές, οι οποίες ε, καταχρώνται των δυνατοτήτων που έχουν σε συγκεκριμένες χώρες. Facebook, πάρτε το Facebook. Το Facebook έχει 30 εκατομμύρια συνδρομητές στη Γαλλία και δεν πληρώνει ούτε ένα ευρώ. Ε, το ίδιο στην Τσεχία, 2-3 εκατομμύρια. Ε, δεν πληρώνει κανένα φόρο. Τώρα εσείς το βρίσκετε κανονικό αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι το είδος του προβλήματος το οποίο προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε. Προφανώς σε μία πρώτη φάση θα υπάρξουν κάποιες χώρες οι οποίες θα έχουν απώλειες φορολογικές λόγω της επιβολής του νέου συστήματος της φορολογικής βάσης. Άλλες χώρες οι οποίες θα κερδίσουν και γι' αυτό ακριβώς προτείνουμε αυτό το Ταμείο Αντιστάθμισης και κάποιοι από εσά είπαν ότι αυτό τους παρουσιάζει ενδιαφέρον, θα ήθελαν όμως περισσότερες διευκρινήσεις. Συνεπώς, πρόκειται για ένα ταμείο το οποίο εγώ θα χαρακτήριζα προσωρινό ταμείο. Θα πρέπει να δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Κάποιοι από εσά το είπαν και οι οικονομολόγοι έχουν κάνει σημαντικές μελέτες επ' αυτού. Όταν μειώνεται η φορολογία αυτό μπορεί να αυξήσει τον πλούτο των φορολογουμένων, διότι είναι προφανές ότι το επίπεδο φορολογίας ε, μειώνεται, οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο θεωρητικά θίγει τα φορολογικά έσοδα. Θα δούμε λοιπόν σε 3, 4, 5 χρόνια ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν και ανάλογα με τα στοιχεία θα κάνουμε τις απαιτούμενες διορθώσεις. Τώρα ένα τελευταίο σημείο σχετικά με τη στάθμιση των κριτηρίων κατανομής. Και εδώ μπορούμε, αν θέλετε, να ρυθμίσουμε κάπως τα πράγματα, ακούγοντας προσεκτικά τα λεγόμενα των μεν και των δε. Θέλουμε εμείς να απαγορεύσουμε τις επιχειρήσεις γραμματοκιβώτια. Θέλουμε ακριβώς να πούμε ότι η κατανομή του φορολογικού βάρους θα πρέπει να λαμβάνει κριτήρια όπως οι πωλήσει, τα ενεργά στοιχεία και το προσωπικό, το ανθρώπινο δυναμικό. Και προτείνουμε εμείς να βάλουμε και τα στοιχεία τα οποία ηλεκτρονικά μπορούν να συλλεγούν τώρα ε, ισότητα των τεσσάρων κριτηρίων ή μπορούμε να τα προσερμόσουμε τα κριτήρια αυτά και το βάρος τους, τη στάθμισή τους για να λάβουμε υπόψη μας ε, κάποιες συγκεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες ή κάποιες συγκεκριμένες χώρες μέλη. Ευχαριστώ όλους όσους πήραν το λόγο. Θα είμαστε μαζί με τον Πολ Τάνκα πολύ προσεκτικοί σε αυτά τα οποία είπατε και θα θέλαμε να συνεχίσουμε τις επισκέψεις της χώρας σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, αλλά θα ήθελα να τελειώσω θυμίζοντας κάποιους αριθμούς. Δεν θα μιλήσω για τα Starbucks, Fiat, Apple, Google. Να πω ότι έχουν κατατεθεί ήδη οι τροπολογίες, θα εξετάσουμε τις τροπολογίες την 6η Νοεμβρίου, θα ψηφίσουμε την 4η Δεκεμβρίου στην ΕΚΟΝ και στην Ολομέλεια τον μήνα Ιανουάριο. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω για την πειθαρχία την οποία επιδείξατε. Νομίζω ότι ήταν επιτυχεστάτη η συνάντησή μας. Πράκεται για θέματα πολύ περίπλοκα. Θα παραμείνουμε όλοι δεκτικοί και θα καταλήξουμε στις επιθυμητές λύσεις. Να κλείσω λοιπόν τη συνεδρίαση λέγοντας ότι η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής ΕΚΟΝ θα είναι στις 16 Οκτωβρίου την τρίτη απογευματινή να ευχαριστήσω όλους. Καλό απόγευμα και ελπίζω να συναντηθούμε σύντομα.